μας. Σήμερα αύριο την Πέμπτη έχετε και την ημερήσια διάταξη, δεν ζητεί κανείς αλλαγή, εγκρίνεται. Στο σημείο 2, οι γλώσσες ε, έχουν προβλεφθεί, γίνεται και αναμετάδοση από το διαδίκτυο για την έγκριση των πρακτικών αυτά που συνηθίζομαι ισχύουν. Ε, εγκρίνονται αν δεν γίνουν ε, αιτήματα για αλλαγές. Πάμε στο 4 απαλλαγή 2017. Έχουμε την Επίτροπο, κυρία Κρέτου, καλώς ήρθατε. Τελευταία φορά, τελευταία φορά είναι μάλλον, δεν το ξέρουμε αυτό, απαλλαγή 2017, προϋπολογισμός της Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς ε, Έχουμε την εισηγητριά μας την κυρία Ινέσα Γιάλα Ζέντερ και έχουμε και εκπροσώπηση ε, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Thank you. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια, κυρία Επίτροπε, αξιότιμα μέλη κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω το κεφάλαιο 6 της ε, ετήσιας έκθεσης του 2017 για την πολιτική συνοχή ως μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτό σχετίζεται με τον υποτομέα 1β του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και καλύπτει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τη διαχείριση της σχετικής δαπάνης από τις DG Regio και Emple. Θα ξεκινήσω την παρουσίασή μου επισημένοντας ότι στον έλεγχό μα ε, για τη δήλωση αξιοπιστίας του 2017 είδαμε ότι η συμμετοχή επηρεάστηκε από διάφορους παράγοντες. Είναι σημαντικό να μην του ξεχνάμε καθώς θα εξετάζουμε τι πληροφορίε που θα σα παρουσιάσω σήμερα. Πρώτον, υπάρχει ένα νέο πλαίσιο ελέγχου και αξιοπιστία. Το νομικό πλαίσιο για το 2014-2020 περιλαμβάνει πολλά νέα στοιχεία. Γεγονό που σημαίνει ότι το επομένων ποσοστό σφάλματο μετά από διορθώσει ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα ή ομάδα επιχειρησιακών προγραμμάτων θα πρέπει να είναι κάτω από το όριο σημαντικότητα του 2% σε ετήσια βάση. Το 2017 ήταν το πρώτο έτος όπου η Κομισιόν δέχτηκε λογαριασμού και καθάρισε δαπάνε που τα κράτη-μέλη είχαν απαιτήσει στο πλαίσιο του νέου αυτού πλαισίου ελέγχου και αξιοπιστία. Δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα ήταν ο περιορισμένο αριθμό λογαριασμών και επενδύσεων που έχουν υποβληθεί το Μάιο του 2017. Η Επιτροπή δέχτηκε λογαριασμού ε, δαπανών από 17 κράτη-μέλη που καλύπτουν μόνο 70 από το σύνολο των 319 επιχειρησιακών προγραμμάτων και δαπανών μόνο 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου. Δεδομένων των κλεισιμάτων της περίοδου 2017-2013, ο πληθυσμός ελέγχου μας καλύπτε μόνο 8 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανών, πολύ λιγότερο από το προηγούμενο έτος που ήταν 36 δισεκατομμύρια για τη δήλωση αξιοπιστίας του 2016 και για το επόμενο έτος που υπολογίζουμε ότι θα είναι 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν έκαναν δαπάνε, αλλά ότι για διάφορου λόγου δεν υπέβαλαν αίτημα επιστροφή αποσμέσεω στην Κομισιόν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η υψηλή αναλογία των δαπανών Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνεχή και ε, Πρωτοβουλία Απασχόληση των Νέων στον ελεγχόμενο πληθυσμό. Κανονικά το στοιχείο αυτό είναι πολύ μικρότερο από το ERDF και το ε, Ταμείο Συνοχή. Αντιστοιχεί στο γεγονό ότι το συνολικό κονδύλιο ESF YEA για τα επιχειρησιακά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020 είναι 26%. Ωστόσο, στον έλεγχο του 2017 η αναλογία των συγχρηματοδοτούμενων δαπανών του Κοινωνικού Ταμείου ε, ανήρχεται στο 48% του πληθυσμού ελέγχου. Ένα άλλο ζήτημα ήταν φέτο ήταν η πρώτη χρονιά που οι, άλλες, ε, που οι ηλεκτρικέ ορχέ υλοποίησαν το νέο πλαίσιο για το 2014-2020. Επιπλέον είχαν ασχοληθούν για πρώτη φορά με τα κλεισίματα τη περίοδου 2007-2013. Το πιο σημαντικό θέμα είναι ότι για την περίοδο 2018-2020 στη σχετική στρατηγική αποφάσισε το ελεκτικό συνέδριο να δει με ένα νέο μάτι το πώς θα ελέγχουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την προστέμενη αξία στη δήλωση αξιοπιστία μας. Ειδικότερα αυτό περιλαμβάνει αυξημένη χρήση της εργασίας άλλων ελεγκτών και των πληροφοριών ε, που παρέχουν οι ενεχόμενοι για την τακτικότητα των δαπανών. Γι' αυτό το σκοπό ε, ο έλεγχος ήταν μια πιλωτική άσκηση το 2017 για τη δήλωση αξιοπιστίας με σκοπό να υποφεληθούμε από το νέο πλαίσιο ελέγχου και αξιοπιστίας για την περίοδο αυτή και να μειώσουμε το διοικητικό φόρτο των τελικών δικαιούχων. Η υλοποίηση του πιλωτικού εγχειρήματο περιλάμβανε την τροποποίηση τη προσέγγιση ελέγχου μα με σκοπό δύο στόχου. Δηλαδή, να συμβάλλουμε στη συνολική δήλωση αξιοπιστία, όπω και στα προηγούμενα έτη και ένα νέο στοιχείο να αξιολογήσουμε το νέο πλαίσιο ελέγχου και αξιοπιστία και το βαθμό στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Αυτό θα μα βοηθήσει να καταλάβουμε στο μέλλον να μπορούμε να αυξήσουμε τη χρήση των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτό και να διευκολύνουμε αυτό ώστε να δούμε πού χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσει. Γι' αυτό το σκοπό ε, κάναμε δειγματοληψία συναλλαγών, τι οποίε εξετάσαμε και τι οποίε είχαν εξετάσει ήδη οι ελεγκτικέ αρχέ των κρατών μελών. Σε σχέση με τον, με τον πρώτο στόχο τη νομιμότητα και τη τακτικότητα, για τον έλεγχο μα εξετάσαμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 217 συναλλαγών που καλύπτουν 51 επιχειρησιακά προγράμματα, 29 επιχειρησιακά προγράμματα από την περίοδο 14-20 και 22 τη περίοδου 7 έω 13. Ελέγξαμε τις συναλλαγές με αναθεώρηση των ληστών ελέγχου των ελεκτικών αρχών και των στοιχείων που είχαν για να τεκμηρώνουν το αποτέλεσμα του δικού του ελεκτικού έργου και των δικών του γνωμοδοτήσεων. Όπου δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα βάσει τη δική του εργασία, ξανακάναμε τον έλεγχο. Σε... Αυτό συνέβη σε 121 τέτοιε συναλλαγέ. Αυτό συμπεριέλαβε 80 επισκέψει επιτόπου σε επίπεδο δικαιούχων. Το 2017 το εκτιμόμενο επίπεδο σφάλματο για το ε, υποτομέα 1β ήταν 3%. Δηλαδή περαιτέρω μείωση σε σχέση με πέρυσι που ήταν 4,8% και το έτο πριν από αυτό που ήταν 5,2%. Οι συνεχεί προσπάθειε όλων των συμμετεχόντων στην ελεγκτική αλυσίδα βοήθησαν να βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Επίση, πρέπει να σημειωθεί ότι το αναφερόμενο εκτιμόμενο επίπεδο σφάλματο είναι για πρώτη φορά χωρίς διορθώσεις. Ε, ουσιαστικά αναφέρεται στα σφάλματα που έχουν εντοπίσει τα κράτη-μέλη, οι ελεκτικέ του αρχέ βασικά. Επιπλέον, όπω αναφέρθηκε πριν, οι διάφοροι παράγοντε επηρέασαν τον έλεγχο τη ε, συνοχή το 2017. Παρότι εξετάσαμε μόνο ε, ήδη ελεγμένε συναλλαγέ, το επίπεδο ασφάλματο που εκτιμήσαμε περιλαμβάνει 36 ποσοτικοποιημένα ασφάλματα που δεν ανείχνευσαν οι ελεκτικέ αρχέ των κρατών μελών. Τα χρηματοοικονομικά μέσα ε, ε, ήταν το μεγαλύτερο μερίδιο ε, στα σφάλματα και ακολουθούμενα από τα μη επιλέξιμα κόστη και τα μη επιλέξιμο ΦΠΑ. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, η χρήση τους αυξάνεται διαρκώς. Αυτό σημαίνει ότι είναι όλο και πιο σημαντικά τα ευρήματά μας σε αυτόν τον περίπλοκο τομέα. Στην περίοδο 2007 έως 2013, Ελέγξαμε χρηματοδοτικά μέσα, κυρίως προς υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και βρήκαμε ότι σε μεγάλο βαθμό 80% είχαν επενδυθεί σε εταιρείε που δεν ήταν μικρομεσαίες επιχειρήσει. Σε μια άλλη περίπτωση βρήκαμε μια ελεγκτική αρχή που δεν είχε νομικό δικαίωμα να πραγματοποιεί επαληθεύσει σε επίπεδο χρηματοδοτικού ενδιαμέσου ε, στο πλαίσιο τη πρωτοβουλία για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και έτσι χρειάστηκε να ξανακάνουμε 30 συναλλαγέ για αυτό το χρηματοδοτικό μέσο και βρήκαμε ότι 9 από αυτέ δεν ήταν επιλέξιμε διότι ο δικαιούχο είτε δεν ήταν μικρομεσαία επιχείρηση ή πραγματοποιούσε μια επιλέξιμη δραστηριότητα. Για το μη επιλέξιμο ΦΠΑ και τα σχετικά προβλήματα, αυτά τα βλέπουμε συχνά στι αιτήσει εκθέσει μα. Ε, στην έκθεση του 2017, Στην δήλωση εξεπιστία, βρήκαμε 10 ε, έργα σε 5 επιχειρησιακά προγράμματα που οι αρχέ των κρατών μελών δήλωσαν ε, επιστρεφόμενο ΦΠΑ ω επιλέξιμη δαπάνη ενώ δεν θα έπρεπε. Το δικαστήριο προετοίμασε μια ταχεία αναθεώρηση των υποθέσεων σε σχέση με το ΦΠΑ η οποία θα δημοσιευτεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Ο δεύτερος ε, στόχος του ελέγχου μας ήταν να εξετάσουμε το νέο πλαίσιο ελέγχου ε, και αξιοπιστίας για την περίοδο 14-20 και το πώς μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό για το μέλλον. Δεδομένου ότι ήταν πιλωτικό το εγχείρημα φέτο, ένα σημαντικό κομμάτι το αφιερώσαμε στην αξιοπιστία, στην αξιολόγησή του. Η δική μα αξιολόγηση του πλαισίου αυτού καλύπτει τι εργασίε των κρατών μελών και των αρχών του που επικύρωσαν τι πληροφορίε που ελαμβάνονταν στα δέσμη ε, εγγράφων που δόθηκαν για την αξιοπιστία και για το κλείσιμο. Εξετάσαμε δηλαδή το έργο των ελεκτικών αρχών των κρατών μελών. Είναι σημαντικό κομμάτι ε, όσον αφορά τι δαπάνε στο πλαίσιο τη ε, συνοχή. Εμεί ελέγξαμε 21 ελεκτικέ αρχέ στην περίοδο 2014-2020 για τα κράτη-μέλη που είχαν υποβάλει τέτοιε δέσμε εγγράφων για την αξιοπιστή ε, ολόγησή μα. Κατέληξε σε διάφορα ευρήματα με ελλείψει όσον αφορά το έργο των ελεκτικών αρχών που περιορίζουν την αξιοπιστία του. Σε 9 από τι 22 δέσμε εγγράφων αξιοπιστία κλεισίματο όπου υπήρχε ε, συντελεστή σφάλματος κάτω του 2% ήταν πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Έπρεπε να είναι πάνω από το όριο σημαντικότητα στην πραγματικότητα. Επίσης εντοπίσαμε διάφορες αδυναμίες όσον αφορά το έργο των ηλεκτρικών αρχών. Αυτές αφορούν την αντιπροσωπευτικότητα των δεγμάτων και το εύρος, στην ποιότητα και την τεκμηρίωση των εργασιών τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις έπρεπε να επαναληφθούν οι συναλλαγέ οι οποίε απέτησαν επιπλέον πόρου του ελεγκτικού συνεδρίου με αποτέλεσμα επιπλέον φόρτο για τον δικαιούχο, επειδή χρειάστηκε να επισκεφθούμε 80 δικαιούχου οι οποίοι είχαν ήδη λάβει την επίσκεψη μια ελεγκτική αρχή. Όσον αφορά το έργο τη Κομισιόν, ο κύριο τη ρόλο στο νέο πλαίσιο είναι να δέχεται ή όχι του λογαριασμού που περιλαμβάνονται στις με γράφων για την εξοπιστία που λαμβάνονται και να διασφαλίσει την κανονικότητα των σχετικών δαπανών. Τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών συνέβαναν στη δήλωση εξοπιστίας του Γενικού Διευθυντή στην ε, αίτηση έκθεση δραστηριοτήτων. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα με το εναπομένον συντελεστή σφάλματο Στην έκθεση αυτή πρώτον υπάρχει πολλά σφάλματα σε αυτή την ετήσια έκθεση, 13 στην DG Regio, με διαφορετικές περιόδους αναφοράς. Οι ετήσιες εκθέσεις του 2017 έχουν πρόβλεψη συντελεστή σφάλματος για τις ε, ε, δηλώσει αξιοπιστία ε, που δεν έχουν ακόμα περάσει από τον πλήρη κύκλο ελέγχων επιπλέον για μια αναλογία των επιχειρηματικών προγραμμάτων που ελέξαμε. Το υπολογιζόμενο, ε, ο υπολογιζόμενο συντελεστή σφάλματο ήταν πάνω από το όριο σημαντικότητα του 2%. Λοιπόν, συνολικά κυρίε και κύριοι, είδαμε διάφορε ελλείψει υπάρχουν εδώ πέρα και συμπεράναμε ότι χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσει, ειδικότερα όσον αφορά το πλαίσιο υλοποίηση από τι ελεκτικέ αρχέ και σε επίπεδο κομισιών. Έτσι, θα συνεχίσουμε με την ίδια ελεκτική προσέγγιση για το 2018. Κάναμε έξι συστάσει με σκοπό να βελτιωθεί η κατάσταση στο μέλλον, τρει από τι οποίε έχει δεχτεί η Κομισιόν, ενώ οι άλλε τρει έχουν γίνει δεκτέ εν μέρη ενώ προφανώ ε, τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δαπανώνται σύμφωνα με του κανόνε, είναι πολύ σημαντικό να έχουν θετική επίδραση όσον αφορά τα αποτελέσματα και τους στόχους. Για τέταρτη, χρονιά φέτος, για τέταρτη φορά φέτο είχαμε ένα ειδικό τμήμα στο κεφαλαίο 6 που αφορούσε τις αποδόσεις, την απόδοση στην πολιτική συνοχή. Αξιολογούμε σχετικά την απόδοση 113 επιχειρηματικών προγραμμάτων που είχαν ολοκληρωθεί τη στιγμή του ελέγχου 56 για την περίοδο 7 έως 13 και 57 για την περίοδο 14 έως 20. Αξιολογήσαμε πρώτα απ' όλα το σχεδιασμό του συστήματο απόδοση και αντιληφθήκαμε ότι ένα σύστημα μέτρηση απόδοση υπήρχε για τα 2 τρίτα των σχεδίων των προγραμμάτων που ελέγξαμε. στι περισσότερε άλλε περιπτώσει δεν είχαν καθοριστεί επαρκεί δείκτε αποτελέσματο σε επίπεδο προγράμματο και ήταν δύσκολο να αξιολογηθεί η συνολική συμβολή ενό έργου στου στόχου ενό συγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματο. Αξιολογήσαμε τι αποδόσει αυτών των 74 έργων για τα οποία είχαν οριστεί και δείκτε αποτελεσμάτων και απόδοση. Αυτό μα βοήθησε να δούμε κατά πόσο τα αποτελέσματα που δήλωναν τα κράτη-μέλη σχετίζονταν ε, με του ε, σχετικού στόχου. Βρήκαμε ότι όλες οι δείκτες ε, που είχαν αναφερθεί ε, τηρούνταν. Για να κλείσω, ελπίζω αυτά τα συμπεράσματα και οι συστάσεις να βοηθήσουν την Επιτροπή σας. Η σημαντικότητα αυτού του τομέα πολιτικής ε, φαίνεται στο γεγονός ότι 7 εκθέσεις έχει ε, εκδώσει το ελεγκτικό συνέδριο για θέματα συνοχής το 2017 και 11 το 2018. Επίση, έχουμε την γνωμοδότηση 6 του 2018 που παρέχει τι δικέ μα απόψει για την πρόταση ενός, για ένα κανονισμό κοινών διατάξεων που θα διέπει το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Θα κλείσω αναγνωρίζοντα ε, καλή συνεργασία και επικοδομητική συνεργασία που έχουμε με την Κομισιόν σε όλη τη διαδικασία. Και τέλο, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Γιάλα Σέντερ για την πολύ χρήσιμη μεταλλαγή απόψεων σε σχέση με αυτή τη διαδικασία απαλλαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Επίτροπος, η κυρία Κρέτσου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Ισηγήτρια, αξιότιμα μέλη, ε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Επιτροπή σας για τη μεγάλη πολιτική στήριξη που παράσχατε όλα αυτά τα χρόνια. Συνεργαστήκαμε και πετύχαμε πολλά. Είμαστε περήφανοι σε ό,τι αφορά την νομιμότητα αλλά και την κανονικότητα. Όπως ξέρετε και όπως ακούσαμε φέτος το ελεγκτικό συνέδριο είδε τις βελτιώσεις για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και στην πολιτική συνοχή βρήκε βελτιώσεις. Για χρόνια είχαμε ε, καθοδική τάση στο ποσοστό σφάλματος. Ελπίζω αυτή η καθοδική τάση να συνεχίσει. Στην αρχή της θητείας μου, της εντολής μου, είχαμε 5,7% ποσοστό σφάλματος. Τώρα πέσαμε στο 4,8%. Πέρσι 4,8% και τώρα 3%. Η πρόοδος ε, οφείλεται σε δύο τινά. Ε, πιο ισχυρό νομικό πλαίσιο και μεγαλύτερη οριμότητα στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Και ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε χρόνο, χρόνο τα προγράμματα, στα προγράμματα γίνονται οι δημοσιονομικές διορθώσεις και η συνεργασία μας με τα κράτη-μέλη αποδίδει. Επίσης, ε, χαίρομαι με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να προσαρμόσει την προσέγγιση ελέγχου. Το πλαίσιο για τον έλεγχο και την αξιοπιστία ενισχύθηκε και μέχρι το 2014-2020 απέδωσε. Τώρα παρακολουθεί όλη την αλυσίδα του ελέγχου και επίσης το ελεγκτικό συνέδριο έλαβε υπόψη και τις διορθώσεις που έχουν ήδη γίνει. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την πρωτοβουλία αυτή, ευθυγραμμιζόμαστε για να μπορούμε να μετράμε και εμείς με το σύστημά μας τα σφάλματα και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε επικαλύψεις των λεκτικών προσπαθειών συνεχίζουμε να επιμένουμε ε, και βασιζόμαστε στα επιτεύγματα. Του χρόνου θα είναι μεγαλύτερες οι δαπάνε και πρέπει να, είμαστε, ε, να επαγρυπνούμε. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες με τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουμε τη λειτουργία των ε, συστημάτων τους όπου χρειάζεται και παρακολουθούμε και πρόσθετα σφάλματα αλλά που θα συνεπάγονται πρόσθετες διορθώσεις αν χρειαστεί. Τώρα θα ήθελα να Κάνουμε έναν απολογισμό που βρισκόμαστε στο κλείσιμο των προηγούμενων προγραμμάτων, εφαρμογή των τωρινών προγραμμάτων, υλοποίηση των προγραμμάτων και πρόταση για, το, για μετά το 2020. Για το κλείσιμο. Τώρα έχουμε προχωρήσει στη διαδικασία πολύ για την περίοδο 2017-2020, προγραμματική περίοδο, και με χαρά θα ακούσαμε ότι το κλείσιμο προχωράει πολύ ταχύτερα από τις οποιαδήποτε άλλη προγραμματική περίοδο. Έχουμε προσωρινό ή ολοκληρωτικό κλείσιμο πάνω από 30 προγράμματα και θα προχωρήσουμε και σε άλλα μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν θα κλείσουμε κανένα πρόγραμμα βέβαια, εκτός και αν έχουμε λογικοφανή αξιοπιστία. Ε, σχετικά με τις δαπάνες. Τα κράτη-μέλη πιστεύουμε ότι έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν και ήταν πολύ σοβαρά διότι εφήρμασαν δημοσιονομικές διορθώσεις στα πακέτα του κλεισίματος που υπευλήθησαν και εμείς από την πλευρά μας είδαμε εντελεχώς την κατάσταση κάθε προγράμματος εφαρμόσαμε τι, τα πρόστιμα και τις δημοσιονομικές ε, διορθώσεις κάθε φορά που υπήρχαν ανοιχτά θέματα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε έτσι. Ε, ε, πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τους ε, εφαρμοστέους κανόνες, μειώθηκε το ποσοστό σφάλματος, επειδή αυτό επιβεβαιώνει τα συστήματα λειτουργούν καλύτερα, έτσι μπορούμε να εστιάσουμε περισσότερο στις επιδόσεις. Οι επιδόσεις πάντοτε ήταν ο στόχος μας και πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε την προστιθέμενη αξία των πολιτικών μας, τον αντίκτυπο των πολιτικών μας και αυτή η χρονιά είναι ιδιαίτερα κρίσιμη πριν από τις ευρωεκλογέ για να δείξουμε και εμείς τι μπορεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική βοήθεια στις περιφερειές μας, στις χώρες μας, στις πόλεις μας και πρέπει και εμείς να παίξουμε το ρόλο μας διευκολύνοντας τις σχετικές συζητήσεις με τους πολίτες και για τους πολίτες. Και πάω στο δεύτερο σημείο. Ε, επιταχύνομαι στην υλοποίηση των τωρινών προγραμμάτων. Η υλοποίηση επιτόπου σαφώς έχει βελτιωθεί και τα το ποσοστό των projects που επιλέγονται είναι παρόμοιο με τις προηγούμενες χρονιές. Περίπου το 70% της χρηματοδότησης είχε δοθεί στα προγράμματα μέχρι τον Νοέμβριο. 366 δις από την πολιτική συνοχή και το Περιφερειακό Ταμείο, 250.000 project. Αυτά είναι επενδύσεις με πολύ καλά στοχοθετημένε, βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων. 250.000 θέσει εργασία θα δημιουργηθούν έτσι πάνω από 4 εκατομμύρια πρόσθετα νοικοκυριά θα καλυφθούν και πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι θα βελτιωθούν από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας. 50 εκατομμύρια πολίτες θα ωφεληθούν από μέτρα ε, πυρόσβεσης. Ε, επίσης, ε, υπήρχαν και άλλα παρεπόμενα ωφέλη από τη βελτιωμένη ρεσιμότητα, καλύτερη διακυβέρνηση των δημοσίων πολιτικών στα κράτη-μέλη, καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον που οδηγεί σε πολιτικές ε, μεταρρυθμίσεις και βελτιώνει την ικανότητα των δημοσίων θεσμικών οργάνων. Η Κομισιόν θέλει πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις και την υλοποίηση επιτόπου. Όλοι πρέπει να παρακολουθούν τα συγκεκριμένα επιτεύγματα των προγραμμάτων με την πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων που υπάρχει. Η πλατφόρμα αυτή δείχνει και τα ε, δημοσιονομικά επιτεύγματα της προηγούμενης ε, περίοδου. Δεν είναι τυχαίο ότι η πλατφόρμα αυτή κέρδισε και ένα βραβείο ευρωπαϊκό, διότι είναι άρτια εις ό,τι αφορά τη δημόσια διοίκηση. Αυτό έγινε το 2017. Πρέπει όμως να ομολογήσουμε ότι η καλή υλοποίηση επιτόπου θα πρέπει να μεταφράζεται 100% και σε σωστή δημοσιονομική ε, οικονομική χρηματοδοτική εκτέλεση. Ε, το επίπεδο απορρόφησης είναι χαμηλότερο φέτος από ό,τι περιμέναμε. Αυτό οφείλεται ε, στο πιο χαλαρό εν συν κανόνα για την αποδέσμευση και έχει να κάνει και με το γενικότερο σύστημα των προκαταβολών ε, που βέβαια υπόκειται σε αυστηρότερους ελέγχους αλλά η χαμηλή απορρόφηση φυσικό είναι να οδηγήσει σε περισσότερες εκκρεμείς δεσμεύσεις σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους. Όμως το ο κανόνας N συν θα αρχίσει να έχει αποτελέσματα για όλα τα προγράμματα φέτος και σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο δεν υπάρχουν παρεκκλήσει. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ την κατάσταση σε κάθε πρόγραμμα και συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να επιταχύνουμε την υλοποίησή του. Κυρίε και κύριοι, από την αρχή τη εντολή μου ε, βοήθησα τα κράτη-μέλη, τι περιφέρειε και τι πόλει ώστε να πάρουν περισσότερα κονδύλια από εμά. Και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό μέχρι την τελευταία μέρα τη εντολή μου. Η πολιτική τη συνοχή είναι πολύ ε, ε, ζωτική ε, πηγή χρηματοδότηση για πολλά κράτη-μέλη. Βοήθησε να αντιμετωπιστεί η χρηματοπιστωτική κρίση και βοηθάει και στην ανάκαμψη. Ε, η καταπολέμηση των περιφερειακών ανισοτήτων είναι ένας στόχος μας. Πολλά κρατημέλη βελτιώθηκαν εδώ παρά την οικονομική κρίση. Αλλά σε εθνικό επίπεδο σημαντικές ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των περιφερειών. Καμιά φορά μεγαλώνουν και οι ανισότητες ή προστίθενται και νέες. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε δύο πρωτοβουλίες βασικές ε, η Catching Up Region, μια πρωτοβουλία και μια άλλη για τη βιομηχανική μετάβαση. Ε, δίνουμε επιτόπια, ε, βοήθηση, υποστήριξη ε, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε περιφέρειας για να ξεπεράσουν τα εμπόδια. Οι πρωτοβουλίες αυτές προχωρούν και εξελίσσονται από την αρχική επιτυχία και είναι βασικό στόχος για το μέλλον. Επίσης έχουμε ειδική task force για καλύτερη υλοποίηση προγραμμάτων τα οποία διέτραχαν κινδύνους. Αυτή η ειδική ομάδα, το task force, έδωσε καλά αποτελέσματα το ποσοστό πρόφηση ήταν καλό, το κλείσιμο βελτιώθηκε και ενδεχόμενες απώλειες αποσοβήθηκαν. Ε, αυτό αναγνωρίζεται, αναγνωρίζεται και στην έκθεση για την απορρόφηση. Η ειδική ομάδα εξακολουθεί να συνεργάζεται με τα προγράμματα που τη χρειάζονται. Ε, πέρα από τις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη και τους δικαιούχους, πολύ νωρίς στην εντολή μου επίστην ότι χρειάζεται περισσότερη απλούστευση. Πήρα την πρωτοβουλία πριν από τρία χρόνια να δημιουργήσω υψηλού επίπεδου ομάδα για την απλούστευση για τους δικαιούχους και οι συστάσεις οδήγησαν σε ένα κανονισμό ε, omnibus και καλύπτουν και τις προτάσεις μας για την περίοδο μετά το 2020. Προτάσεις για το μέλλον τώρα. Εμείς δράσαμε αντιμετωπίζοντας ε, τις ανάγκες των κρατών μελών και των δικαιούχων. Ε, θέλουμε να κάνουμε πάλι ελκυστική την πολιτική μας, ε, λιγότερο επιρρεπή σε σφάλματα. Τώρα ο κανονισμός πολυνομοσχέδιο, αν θέλετε, το Omnibus ισχύει. Ε, πρέπει να αναλάβουν ε, δράση στα κράτη-μέλη, να ε, αντλήσουν ωφέλη από την απλούστευση και να επιταχύνουν την υλοποίηση επιτόπου. Στις προτάσεις μετά το 2020 που παρουσιάστηκαν το Μάιο κάναμε και άλλες απλουστεύσει. Με 373 δι προπολογισμό μετά το 2020 η πολιτική συνοχή είναι ένας βασικός ε, επενδυτικό μηχανισμός, συνενώνει την Ένωση και φέρνει πιο κοντά την Ένωση στου πολίτες. Οι προτάσεις μας δημιούργησαν και ένα ε, μενού, ένα μείγμα πέντε πολιτικών ε, ε, για να είναι πιο έξυπνες, η Ευρώπη να είναι πιο κοινωνική, πιο ενωμένη, πιο πράσινη. Θέλουμε έτσι να έχουμε έναν έντονο προσανατολισμό προς τις αποδόσεις. Θέλουμε να έχουμε πρόοδο σε όλα αυτά. Επίση. έχουμε βελτιωμένε συνδέσει με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που θέτει τις προτεραιότητες για την πολιτική συνοχή. Και θέλουμε η εφαρμογή να επιταχυνθεί. Ε, πρέπει να είναι ομαλέ οι μεταβάσει μεταξύ προγραμματικών περιόδων, ε, να βελτιωθεί το σύστημα υλοποίηση και να χρησιμοποιηθεί ω πρότυπο. Ε, χρειάζεται πιο αυστηρή δημοσιονομική διαχείριση με τον κανόνα νησιν 2 και λιγότερες προκαταβολές από την Ένωση. Έχουμε μειώσει τη γραφειοκρατία, μειώσαμε τους πολύ σύνθετους κανόνες, εναρμονίσαμε κανόνες ε, σε όλα τα ταμεία και αυτό είναι μεγάλο βήμα μπροστά προς την απλούστευση για τους δικαιούχους και τις αρχές ε, τις προγραμματικές. Έχουμε περίπου 80 μέτρα απλούστευσης ε, στις προτάσεις και ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Ε, για τη διαχείριση και τον έλεγχο έχουμε ισορροπημένη πρόταση για σημαντικές απλουστεύσεις, ε, λιγότερο φόρτο και ελέγχου και έχουμε ε, στιβαρό σύστημα αξιοπιστίας. με τις απαραίτητες επαληθεύσεις εγκρίσεις. θέλουμε θέλω με αναλογικούς ελέγχους στο σύστημα, με καλά αποτελέσματα. Αυτές οι απλουστεύσεις θα βοηθήσουν τους δικαιούχους να επικεντρωθούν περισσότερο στην υλοποίηση επιτόπου. Αγαπητά μέλη, με τις προτάσεις μετά το 2020, αυτές που παρουσιάσαμε, η πολιτική συνοχής θα μπει στη νέα προγραμματική περίοδο ως καλύτερη, πιο σύγχρονη, πιο ευέλικτη πολιτική. Η πολιτική συνοχή θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των περιφερειών, των πόλεων και των τοπικών κοινοτήτων μας. Θέλουμε η πολιτική να συμβάλλει σε μια Ευρώπη που συνδέει τους λαούς, τους, τις περιφέρειες, που ενδυναμώνει τους ανθρώπους για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικέ προκλήσεις, που τους προστατεύει η πολιτική αυτή πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις για το νομοθετικό πακέτο, τη νομοθετική δέσμη. Χαίρομαι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε ταχύτατα στην αξιολόγηση της πρότασης, καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις, απευθύνω έκκληση σε όλα τα θεσμικά όργανα, κυρίως στο Συμβούλιο, να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσουμε τι συμπληρωματικότητε και τι απλουστεύσει. Στου επόμενου μήνε θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν ώστε η δυναμική αυτή να συνεχιστεί στο έργο με τον συνομοθέτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξή σα. Είσαστε αυστηροί, αλλά πολύ επικοδομητικοί. Και πραγματικά το εκτιμώ αυτό το πράγμα, διότι μαζί μας δημιουργείται πιο αποτελεσματική πολιτική συνοχή, μια πολιτική που δίνει τη θέμενη αξία, πολιτικές που δίνουν αποτελέσματα για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους πολίτες και βέβαια ε, σας ευχαριστώ σε αυτό το σημείο για την ε, προσοχή και περιμένω ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Η εισηγήτρια, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και τον κύριο Μέρφυ για την παρουσίαση που έκανε. Είναι αλήθεια πως και για το ελεγκτικό συνέδριο η χρονιά αυτή ήταν δύσκολη. Με ποια έννοια. Χρειάστηκε και αυτοί να θέσουν σε ισχύ μία σειρά από νέα σχέδια για το πώς θα κάνουν τους ελέγχους, και για το πώς θα αξιολογούν τις εκθέσεις και τις ε, έρευνες που κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Κρέτου, με την οποία πάντα συνεργαζόμαστε και θα την παρακαλούσω θα την παρακαλούσα να μας στείλει γραπτά την παρουσίαση που έκανε, γιατί την βρήκαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το μέλλον πλησιάζει το 2019 που είναι ένα κομβικό σημείο γιατί κλείνει ένας κύκλος με τις διαπραγματεύσεις που είναι περίπλοκες για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές και με άλλες διαπραγματεύσεις πολύ σημαντικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Brexit και τις ευρωεκλογέ. και όσα αυτά σημαίνουν εν ώψη ε, τις θέσεις εφαρμογή των μελλοντικών προγραμμάτων. Και θα ήθελα και να σας συγχαρώ γιατί το ελεγκτικό συνέδριο αναγνώρισε σαφέστατα πως έχουμε μεγάλη βελτίωση ε, στο ποσοστό σφάλματος και νομίζω ότι είναι σωστό να αναγνωρίσουμε ότι μετά από τόσα πολλά χρόνια που δουλέψαμε, που υπενθυμίσαμε, που επιστρέψαμε και χτίσαμε νέους τρόπους συνεργασίας, εργασίας, έτσι ώστε όλες οι αρχές, σε όλη την αλυσίδα διεύθυνσης για τα διαστοτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο από τη βάση που είναι ο τελικός δικαιούχος μέχρι και την κορυφή που είναι η Επίτροπος να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και νομίζω πρέπει να αναγνωρίσουμε και τη δική σας προσωπική συμβολή που ήταν πολύ σημαντική για το γεγονός πως το Ελληνικό Συνέδριο αναγνωρίζει πως υπάρχει μια τάση μείωσης των σφαλμάτων και των προβλημάτων σε επίπεδο διαχείρισης και κυρίως συνδιαχείρισης, γιατί υπάρχουν όλες οι task force και όλα τα κράτη-μέλη με τις σχετικές αρχές, οντότητες, τοπικές αρχές, περιφερειακές αρχές, δικαιούχους. Όλα αυτά λοιπόν ε, καρποφόρησαν. Βεβαίω έχουμε προβλήματα, μα είναι τόσο μεγάλο το ύψο του προπολογισμού που θα ήταν αδιανόητο να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα και κάποιο σφάλμα κάπου. Αλλά πρέπει να σα πω πω εμείς κινούμαστε ε, προς τη σωστή κατεύθυνση και και αυτό είναι η άμεση διαχείριση, κάτι το οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε φέτος, μια και στην άμεση διαχείριση έχουμε εντοπίσει και εκεί αρκετά προβληματάκια. Να σας πω λοιπόν πως φέτος που το ελεγκτικό συνέδριο και εσείς αναγνωρίσατε πως είναι ένα μεταβατικό έτος, γιατί πρέπει να κλείσουμε την προηγούμενη περίοδο με τα προγράμματα, με τις ανακτήσεις, με τα προβλήματα στα οποία θα πρέπει να εντοπίσουμε αν έφτασε στους τελικούς αποδέκτες και επίσης παράλληλα με την έναρξη της επόμενης ε, προγραμματικής περίοδου ε, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ήδη μας είπατε πως για το 14-20 έχουμε φτάσει στη μέση και έχουμε τουλάχιστον το 1 τρίτο των ποσών που έχουν εκταμιευθεί όμως ένα από τα στοιχεία που εντόπισε το ελεγκτικό συνέδριο και το οποίο θίξατε κι εσείς πολλές φορές, γιατί δεν είναι δικό σας πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εσάς αφορά περισσότερο τα διαφορετικά ταμεία, είναι η απορρόφηση. Είχαμε τεράστιες καθυστερήσεις. Το είχαμε μιλήσει, το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν. Ο διορισμός των εθνικών αρχών, για παράδειγμα, που καθυστέρησε πάρα πολύ να τεθεί σε ισχύ. Δεύτερον, το στοιχείο ευελιξία που είναι ο κανόνα του συν 3 που οδήγησε μια χαλάρωση σε, κάποιες, ε, σε επίπεδο κάποιων αρχών τη στιγμή της ε, εκταμίευσης των πληρωμών γιατί η κρίση δημιούργησε και προβλήματα ρευστότητα και νομίζω ότι εσείς θα μπορούσατε να μας απαντήσετε στο εξή. Με όλα αυτά τα οποία βάλατε εσείς σε ισχύ και τη λύση που είναι να μην έχουμε νησιν τρία πια, αλλά νησιν 2, αυτά φτάνουν. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη από την απάντηση που λάβαμε στο ερώτημα αυτό. Δηλαδή, ποια είναι τα αίτια για τη μία απορρόφηση, γιατί υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι. Κάποια κράτη-μέλη ε, που δεν μπορούν και χρειάζονται τεχνική βοήθεια. Υπάρχουν άλλα που δεν έχουν ε, συγχρηματοδότηση. Το είπε το ελεγκτικό συνέδριο. γιατί έχουν προβλήματα δημοσιονομικά ε, και ένα σώρο ακόμα. Και αυτό το ρωτάμε και απευθυνόμαστε και σε εσά και στο ελεγκτικό συνέδριο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε σε βάθο ποια είναι τα πραγματικά αίτια αυτών των τεράστιων καθυστερήσεων που καμιά φορά είναι μη θελημένε. Οι, οι περιφερειακές αρχές πολλές φορές οι τοπικέ αρχέ δεν τα καταφέρνουν αλλά υπάρχουν και κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε γιατί αυτή τη στιγμή Είμαστε σε ένα εργοτάξιο για να το χαρακτηρίσω έτσι στο οποίο θα χρειαστεί να σκάψουμε πιο βαθιά για να θεμελιώσουμε αυτό που θέλουμε. Γιατί με την καθυστέρηση στην απορρόφηση, το λέει και το ελεγκτικό συνέδριο, τελικά έχουμε τόσες πολλές δεσμεύσεις πληρωμών που θα οδηγηθούμε στο εξή. Τη στιγμή της πραγματικής πληρωμής στο τέλος του κύκλου 14-20 τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί εκεί θα πρέπει να διαπραγματευτούμε τον επόμενο και καλό θα είναι να μην έχουμε όλες αυτές τις πληρωμέ σε εκκρεμότητα ή σε αγκύλες ή σε παρένθεση. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε και να το λύσουμε. Και τέλος θα ήθελα να εντοπίσω ε, ένα ακόμα πρόβλημα που είναι το ποσοστό σφάλματος. Εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, το λέει και το Ελεγκτικό Συνέδριο, το λένε και οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να εντοπίσουμε ακριβώς το σημείο, τη χρυσή τομή, όπου ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εμπλουτίζεται με διάφορα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το τα ποσά των ανακτήσεων. Γιατί με τις καθυστερίες που αντιμετωπίζουμε και με την κατάσταση που έχουμε επιτόπου έχουν πολλαπλασιαστεί οι εκθέσεις και των γενικών διευθύνσεων και των εσωτερικών ελέγχων συν των όσων λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη όπου έχουμε μία πληθώρα ποσοστών σφάλματο που καμιά φορά είναι αντιφατικά μεταξύ του κιόλα που μας δυσκολεύουν πάρα πολύ και δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τι γίνεται γιατί ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή είναι δυναμικό, αλλά θα πρέπει κάθε έτο να μπορούμε να εξηγήσουμε ε, στον ευρωπαϊκό πολίτη και στου δικαιούχου τι ακριβώ κάνουμε και τι ακριβώ εφαρμόζουμε, χωρί να δημιουργούνται μεγάλα ερωτηματικά ε, για το τι συμβαίνει με τον προϋπολογισμό μας. Και τέλος, εγώ σας συγχαίρω. Τα αποτελέσματα στη συνοχή είναι αυτά τα οποία πιο πολύ θετική αναγνώριση έτυχαν από το ελεγκτικό συνέδριο. Αλλά δεν έχουμε ακόμα αξιόπιστου δείκτε, έτσι ώστε να μπορούμε να τα μετρήσουμε όλα αυτά, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Και αυτό λοιπόν ε, θα μείνει για το μέλλον. Σίγουρα και οι συνάδελφοι θα προσθέσουν κάτι. Αν φτάσουμε στο τέλος και δεν τα έχουν πει όλα, θα πάρω και πάλι το λόγο. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Συγήτρια. για τα πολύ θετικά σας ε, σχόλια τόσο όσον αφορά τη δουλειά του Ελεκτικού συνεδρίου όσο και όσον αφορά τη δουλειά της Κομισιόν. Είμαστε σε ιδιαίτερες εποχές, ε, σε, όπως είπατε. Έχουμε περίπλοκες διαπραγματεύσεις για το Brexit, για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας απαντήσω όσον αφορά τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται. Αυτό που μας ενισχύει όλους όπως είπα, η διαδικασία εφαρμογής προχωρά κανονικά. Το ποσοστό επιλογής των προγραμμάτων έχει φτάσει στο 69%. Τα συνολικά κονδύλια για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 14-20. Αυτό αντιπροσωπεύει το 2 τρίτα του συνόλου των ποσών που έχουν δοθεί. Δυστυχώς η Κομισιόν Ε, δεν έχει να το 20% τα μέσα πληρωμών που έχουν δηλωθεί είναι περίπου στο 17%. Βρισκόμαστε σε διαρκή διάλογο με τα κράτη-μέλη για τη βελτίωση της κατάστασης. Παρακολουθούμε στενά τα προγράμματα που θεωρούνται υψηλής επικινδυνότητας και φυσικά Θέλουμε να επιταχύνουμε την αποδέσμευση και την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τα τελευταία χρόνια, πιστεύω, η Κομισιόν έχει υποστηρίξει σημαντικά όλα τα κράτη-μέλη, ειδικότερα μέσω τεχνικής ε, υποστήριξης, ε, υποστήριξης ε, για τη συνδιαλλαγή. Έχουμε στείλει εμπρογνώμονες στα κράτη-μέλη στις περιφέρειες, κάνοντας προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις, να επιλύσουμε τα προβλήματα του συστήματος που καθυστερούν ε, την υλοποίηση και να επιταχύνουμε την υλοποίηση. Οι υπηρεσίε μα είναι διαρκώς ε, στη διάθεση των κρατών μελών. Δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω όσον αφορά το, τα αποτελέσματα για το οποία έχουν δεσμευτεί τα κράτη-μέλη για αυτή την προγραμματική περίοδο. Ήθελα τώρα να σας πω ότι κατά την άποψή μου υπάρχουν κάποιοι λόγοι που έχουν επιβραδύνει τις, απο, τις απορροφήσεις βάσει συζητήσεων που έκανα με δικαιούχους. Τα κράτη χρειάζονται περισσότερο χρόνο μερικές φορές για να καθορίσουν τις αρχές διαχείρισης και ελέγχου. Ξέρετε πολύ καλά ότι στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά προγράμματα έχουμε καθορίσει σαφή κριτήρια ώστε να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούμε να υπολογίζουμε σε αυτά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Γι' αυτό το λόγο ορισμένοι χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να τα υλοποιήσουν αυτά τα καινούργια όργανα αλλά και για να τηρήσουν ε, την ε, εξαντερεσιμότητα. Αυτό, αυτά ήταν απαραίτητα για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ήταν απαραίτητες σε διάφορους τομείς, σε πολλά κράτη-μέλη. Επίση, όπως είπα, τα ποσοστά ε, προχρηματοδότησης είναι πολύ ψηλά κατά την απόψη μα. Ο κανόνα νήσιν 3 όσον αφορά τι δεσμεύσει, ε, τις αναλήψεις υποχρεώσεων, και το υψηλό ποσοστό το υψηλό ποσοστό λοιπόν προχρηματοδότηση και ο κανόνα ε, νήσιν 3 δεν βοήθησαν να ασκηθεί πίεση στα κράτη-μέλη για να τηθούν πληρωμέ στον κανονισμό έχουμε προβλέψει αυτή τη διάταξη της ε, καθαρής διόρθωσης. Αυτό δείξε σε ανησυχία των εθνικών αρχών, διότι μπορεί να υπάρξει αναστολή κάποιων κονδυλίων ή ε, προαναστολή κάποιων κονδυλίων εάν δεν έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες για να έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι αεραγκαίοι έλεγχοι πριν από την υποβολή των ε, δαπανών προς πληρωμή. Κατά την άποψή μου, ε, ένα άλλο λόγο για τι καθυστερήσει ήταν η καθυστερημένη υιοθέτηση αυτή τη νομοθεσία. Ε, για πολύ καιρό δεν υπήρχε σαφή θέση. Υπήρξαν καθυστερήσει όσον αφορά το κλείσιμο των προγραμμάτων 2007-2014 και μετά καθυστέρησαν να ξεκινήσουν τα προγράμματα τη περίοδου 14-20. Αλλά θεωρώ ότι η Κομισιόν έχει αποκομίσει όλα τα μαθήματα που έπρεπε. Γι' αυτό το λόγο για την επόμενη προγραμματική περίοδο προτείνουμε να πλουστευτούν ριζικά οι κανονισμοί με πιο ομαλή μετάβαση από τη μια δημοσιονομική περίοδο στην άλλη για την επόμενη γενιά προγραμμάτων. Πρόκειται για ένα κοινό εγχείρημα, μια κοινή προσπάθεια που θα πρέπει να κάνουμε μαζί ώστε να επιταχύνεται η υλοποίηση επιτόπου. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε στα κράτη-μέλη ότι ε, αυτή η πολιτική συνοχής παράγει απτά αποτελέσματα. Ναι, φυσικά ενίοτε χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο μέχρι να γίνουν ορατά τα αποτελέσματα. Κάποια προγράμματα εκτείνονται σε περισσότερες από μία προγραμματικές περίοδου και τα αποτελέσματα δεν είναι ορατά παρά χρόνια αργότερα. Αλλά πιστεύω ότι στο σύνολο Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά με εσά, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το Ελεγκτικό Συνέδριο, με τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να βρούμε την καλύτερη δυνατή ισορροπία. Είτε μεταξύ απλούστευση ε, των κανονισμών, ε, είτε και για τη διασφάλιση των αποτελεσματικών ελέγχων, ώστε τα χρήματα των φορολογουμένων να δαπανώνται υπέρ του συμφέροντος των πολιτών και βελτιστοποιώντας τα αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Ευχαριστώ. Ναι, τώρα. Να πούμε ορισμένα πράγματα. Ε, ξέρω ότι είναι πλήρης έτσι όπως είναι η συνολική μας προσέγγιση και πολιτική. Το ελεγκτικό συνέδριο ε, άλλωστε ισχυρίζεται ότι οι στόχοι δεν επετεύχθησαν πλήρως. Τι πετυχαίνει η πολιτική σύνοχης, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. δίνονται πολλά χρήματα, πολλά στα κράτη-μέλη. Σίγουρα έχουν τα χρήματα αυτά αποτέλεσμα. Θα ήταν άσχημο αν δεν συνέβαινε αυτό, αλλά δεν πρέπει να βελτιωθούμε. Δεν πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για την ε, μεγέθυνση, την ανάπτυξη, την ε, ανάπτυξη των περιφερειών, τη μείωση ανισοτήτων μεταξύ τους. Η διαφορά και οι ανισότητες έχουν μεγαλώσει, μάλλον παρά μικρύνει, γιατί το τα κονδύλια είναι ένα μόνο μέσον. Αν τα κράτη-μέλη δεν ε, χρησιμοποιούν τα κονδύλια από τις Βρυξέλλες για να στηρίξουν εθνικά μέτρα, τότε δεν πετυχαίνουν. Ε, γι' αυτά θέλω να μιλήσω, τη στήριξη των εθνικών μέτρων και να ρωτήσω σε ποιο βαθμό συνδέονται τα κονδύλια με την ανάπτυξη και την απασχόληση και τη δημιουργία οικονομικών δομών. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω αυτό. Είναι μια ερώτηση γενικής αξιολόγησης και βέβαια μπορούμε να μπούμε και σε λεπτομέρειες που αφορούν το ένα ή το άλλο κράτος μέλος. Τα παραδείγματα είναι πολύ σημαντικά. Ε, τώρα, η αργή πολυ σημαντικα τωρα η αργη διεκπαιρεωση Ε, δεν είναι ότι ε, αρχίζουμε αργά και τελειώνουμε αργά. Είναι ότι όλο και περισσότερο αποκλίνουμε από το στόχο της εδαφικής συνοχής. Το ελεγκτικό συνέδριο λέει για 70 δέσμες και 2,5 δις ευρώ. Δεν είναι πολλά. Ακόμα υπολοιπόμεθα πολύ, περισσότερο από ποτέ. Τι κινδύνους αντιμετωπίζουμε με αυτήν την ταχεία, την βραδία, συγγνώμη, υλοποίηση. Και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Πώς βλέπετε τους κινδύνους της βραδίας υλοποίησης. Ο, ο, ο πολιτικός μας στόχος έτσι δεν αμφισβητείται συνολικά. Επίσης, ε, τα μέσα ε, χρηματοδοτικού ε, ανασχεδιασμού. Το συνέδριο λέει ότι λιγότερο από 10% του financial engineering έχουν φτάσει στον τελικό δικαιούχο. Και εδώ έχουμε πρόβλημα, κυρία Επίτροπε. Τι κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Αυτή είναι η τρίτη μου ερώτηση. Τέταρτη ερώτηση. Κάποια ανησυχητικά ζητήματα, δηλαδή συγκρούσεις συμφερόντων. Στον έλεγχο προϋπολογισμών και ευχαριστώ τη Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο για την καλή μας συνεργασία. Μπορούμε έτσι να εντοπίζουμε ε, συγκρούσεις συμφερόντων άνθρωποι δηλαδή πλούσιοι που κατεβαίνουν και στην πολιτική ή ε, ε, σε άλλα κράτη μόνο οι μέτεροι έχουν πρόσβαση στα κονδύλια ή άλλοι βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν τα κονδύλια για να ανασταλεί η ελεύθερη λειτουργία του ανταγωνισμού. Υπάρχουν και τέτοια κράτη-μέλη βλέπουμε καινούριε εξελίξεις στα κράτη-μέλη γιατί πολλές φορές και τα κονδυλία χρησιμοποιούνται με λάθος τρόπο. Ε, πώς θα αντιμετωπίσετε και τη σωστή χρήση των κονδυλίων. Και τέλος το θέμα της αξιοπιστίας των διαχειριστικών αρχών. Αυτό είναι σαν κόκκινη κλωστή σε όλη την έκθεση διαχείρισης. Πώς μπορούμε να φροντίσουμε ώστε οι καλές δηλώσεις, οι μεγάλες ε, βελτιώσεις ε, θα μας οδηγήσουν σε αξιοπιστία, δηλαδή να έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές διαχείρισης. Ε, πολλές φορές οι αρχές διαχείρισης ε, έχουν και ίδιες συγκρούσεις συμφερόντων και αυτές οι συγκρούσεις συμφερόντων είναι ένα σφάλμα συστημικό και ένα πρόβλημα συστημικό. Πώς θα αντιμετωπίζετε? Μπορούμε να βασιστούμε ότι θα λυθούν αυτά. Δεν θέλω να μου ε, εξηγήσετε το σύστημα ελέγχου, το, δεν περιμένω κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχουν τόσα προβλήματα διαχείρισης και στην αλυσίδα ελέγχου και το ζήτημα είναι αν θα είχε νόημα η Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο θα μπορούσε να εξετάσει τα προγράμματα ένα προς ένα μεταξύ άλλων και όχι σε επίπεδο γενικότερης λειτουργίας συστήματος. Και τώρα η συνάδελφος Λαμπαγιώβα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί επίτροπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη δουλειά που έχετε κάνει και πρέπει να σας πω πως είναι πολύ λεπτομερής οι απαντήσει που δίνεται. Κάνει όλο και καλύτερη δουλειά στι γραπτέ τη απαντήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλέ φορέ. δεν χρειάζεται καν να ζητήσουμε επιπλέον εξηγήσει γιατί είναι τόσο λεπτομερεί οι απαντήσει σα. Και σα ευχαριστώ για τι προσπάθειες που έχετε κάνει για την απλούστευση. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη δουλειά που κάνουμε και δεν έχει να κάνει μόνο με το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και με τι προσθε... προτάσεις που κάνετε για την κατάργηση ρυθμίσεων στο μέλλον. Για μένα αυτή η μείωση στα ποσοστά ασφάλματος συνδυάζεται απόλυτα με την απλούστευση, όπως επίσης και με τα διδάγματα από το παρελθόν. Και έχω ένα φιλοσοφικό περισσότερο ερώτημα που θα ήθελα να σας απευθύνω, αλλά θα ήθελα να δούμε μαζί τι μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον. Γιατί θέλω να μου πείτε τι μορφή θα μπορούσε να έχει η μελλοντική ε, απλούστευση και πώς μπορούμε να μειώσουμε τον νομοθετικό υπερπτηματισμό των κρατών μελών στα πλαίσια του επόμενου δημοσιονομικού ε, πλαισίου και της αιρεσιμότητας. Γίνεται αυτό, απλούσταση παρόλη την αιρεσιμότητα ή μέσω αυτής. Επίσης για τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Τα στοιχεία βασίζονται στις δηλώσεις από τα μεμονωμένα project τα οποία έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στα project αυτά βλέπουμε να αλλάζουν κάποια στοιχεία, για παράδειγμα το επίπεδο χρηματοδότησης, τα αποτελέσματα, τα παραδοτέα. Σας ρωτώ λοιπόν το εξή. Εσείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς αξιολογείτε τα κράτη-μέλη. Ε, με τις δηλώσεις επιτυχίες και με τους δείκτες προβλέψεων. Τα ελέγχετε, αξιολογείτε τα στοιχεία αυτά. Δηλαδή βλέπετε αν είναι σωστά αυτά που δηλώνουν τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Στάς. Όπως και η Μαρτίνα, σας ευχαριστώ πολύ και σας και τις υπηρεσίες σας για τις πολύ λεπτομερείς και αναλυτικές απαντήσεις που μας δώσατε, γιατί μας βοηθήσατε πολύ με τις απαντήσεις σας. Μια ερώτηση που έχει σχέση με αυτά που είπε η κυρία Γκράσλα. Ε, πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ πολιτικών και η, της ιδέας της ε, πληρωμής μεγάλων κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μπάμπιτς, ο Πρωθυπουργό στη Τσεχία, ε, απάντησε ερωτήσεις σχετικά. Θέλω όμως να τα δούμε πιο ξεκαθαρά τα πράγματα. Να Δούμε την πρόσφατη ιστορία και τι έγινε τελευταία. Ε, αρχίζουμε να κάνουμε ερωτήσεις. Νομίζω αυτό έγινε μέσα Σεπτεμβρίου. Μιλήσαμε με τον Επίτροπο Τίνγκερ και είχε πει εκείνος τότε ότι ναι όλα αυτά τα παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Υπήρξε καταγγελία από την Transparency International γιατί κατά της ε, τσεχικής δημοκρατίας θα συνεργαστούμε πολύ και οι γενικές διευθύνσεις ε, Agri, Reggie, Emplo κλπ. Να δούμε τι γίνεται. Ε, Καθησυχάσαμε λίγο, αλλά τέλος Οκτωβρίου ήρθε ο Επίτροπος Χόγκαν, ε, στο Στρασβούργο έγινε αυτό, και ο Επίτροπος Χόγκαν επιβεβαίωσε ότι όντως γίνεται κοινή έρευνα, έτσι την ονόμασε, μεταξύ δηλαδή των τεσσάρων γενικών διευθύνσεων. Οι τέσσερις μαζί κάνουν κοινή έρευνα. Και τώρα στην απάντησή σας, Επίτροπε, στην ε, πάλι 34 ή 35 είπατε ότι δεν μπαίνει θέμα κοινή έρευνα, αν κατάλαβα καλά, αλλά υπάρχει καταγγελία από τη διεθνή διαφάνεια κατά της τσεχικής δημοκρατίας. Και ε, το κόμμα των πειρατών, γιατί και αυτοί έστειλαν 10 έγγραφα, για, και που μιλούν για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Και η απάντησή σας είναι ότι η συνήθιση, η τακτική διαδικασία έχει αρχίσει ε, για να αντιμετωπιστεί αυτή η επίσημη καταγγελία. Αυτή είναι η απάντησή σας στην ερώτηση 35. Και από άλλον πήραμε παρόμοια απάντηση και μου κάνει εντύπωση. Και ανησυχώ, γιατί δεν είναι συνήθις υπόθεση αυτή. Είναι πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ Πρωθυπουργού και μιας εταιρεία που παίρνει πολλές επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι συνθισμένα πράγματα αυτά καθημερινά. Και αν γίνεται αυτό, τότε παραβιάζεται ο δημοσιονομικός κανονισμός. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ και εσά και τις υπηρεσίες σας γιατί ζητήσατε τεκμηρίωση, στοιχεία, θέλατε πλήρη στοιχεία και επιμείνατε σε αυτά και νομίζω ότι η Γενική Διεύθυνση Ρέτζη ε, τα χειρίζεται καλά. Λέτε ότι προσπαθείτε να φωτίσετε τα στοιχεία της υπόθεσης και κάνετε έρευνα. Στην απάντησή σας όμως λέτε ότι τα κράτη-μέλη τα ίδια έχουν την κορυφαία ευθύνη ή την απότατη ευθύνη για να εφαρμόσουν όλα τα μέτρα ελέγχουν και να δουν αν τα προγράμματα εφαρμόστηκαν και υλοποιήθηκαν σωστά σε σχέση με την κοινή διαχείριση. Αλλά όταν υπάρχει τέτοιου είδους καταγγελία, τότε το κράτος μέλος πρέπει να δει αν έγιναν σωστά τα πράγματα, αλλά το κράτος μέλος έχει ηγέτη έναν ύποπτο. Έναν μεταξύ των υπόπτων για σύγκρουση συμφερόντων. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Ε, λοιπόν, θα γίνει έρευνα. Κυρία Επίτροπε, αν γίνει πρέπει να γίνει σύντονα, συντονισμένα, γιατί δεν είναι συνήθις η καταγγελία. Είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό και περιμένω την απάντησή σας αυτό. Είπατε επίσης ότι και μοιάζει με τον κύριο Σάτλμαϊρ αυτό που λέτε, ότι θα μας δώσετε, θέλετε περισσότερο χρόνο για να μας δώσετε αποτελέσματα. Τι γίνεται με τις διάφορες φάσεις της έρευνας. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, ε, καλό είναι να ενημερωνόμαστε αν ε, λαμβάνετε μια απόφαση, ε, θα πρέπει να ξέρουμε. Και κλεισμένο των θυρών, αλλά με ενημέρωση. Και μετά από δυόμισι μήνες δεν είναι μόνο το θέμα της πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων με τον Πρωθυπουργό Μπάμπιτς, αλλά υπάρχει και σύγκρουση συμφερόντων με τον Τσέχο ε, Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Τόμας. Τόμας, το γνωρίζετε, άρχισε να γίνεται έρευνα και για αυτό το θέμα από εσά και τις υπηρεσίες σας. Θα το εξετάσετε, θα δείτε αυτές τις ε, καταγγελίες, τι έχει γίνει ή μήπω τρέχει ήδη έρευνα για αυτό το θέμα. Τέλος, ε, ε, τα διακυβεύματα είναι περισσότερα εδώ. Πρέπει να ε, μπει η Όλαφ στην υπόθεση αυτή. Είχατε επαφές με την Όλαφ ή απλώς αφήνετε τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους. Έχουμε και τρεις ακόμα βουλευτές ε, για να τελειώσουμε και τους σκιώδεις. Η κυρία Κρέτσου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε πολλές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα κυρία Πρόεδρε. Ολοκλήρη η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και εσείς η ίδια με την αυστηρότητα μας επιβάλλατε μεγάλη γρήγορση. Φυσικά αυτό είναι ο κοινός μας στόχος, ανέκαθεν υπήρξε. Θέλουμε οι επιδόσεις ε, υψηλές επιδόσεις να χαρακτηρίζουν ε, την περίοδο 14-20. Και όπως είπα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πιο εξελιγμένο σύστημα σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Θα έλεγα μάλιστα ότι πρόκειται για ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα που έχουμε στη διάθεσή μας σε θέματα διαχείρισης και ελέγχου από όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε που, χρησιμοποιούν ε, τα, που χρησιμοποιούνται για τα κοινωτικά κονδύλια. Όπως είπατε και πολύ σωστά μάλιστα, κάποιες φορές κάποια πράγματα μας ανησυχούν. Ε, το κατά πόσο μπορούμε να βασιστούμε στη διαχείριση και στον έλεγχο των εθνικών αρχών. Ε, γι' αυτό το λόγο οι εργασίες της DG Regio, όπως ξέρετε, είναι περιορισμένος και ε, επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε ορισμένα στοιχεία. Επαληθεύουμε κατά πόσο τα στοιχεία που λαμβάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σωστά πραγματικά ε, και αν μπορούμε πραγματικά να βασιστούμε σε αυτά. Ε, υπάρχει λοιπόν, εκφράζεται αυτή η ανάγκη λογική παρέμβαση σε κάθε πρόγραμμα εντό του κανονισμού και στη συνέχεια η έκθεση αποτελεσμάτων ε, έχει παγιωθεί. Το 2019 λοιπόν προτείνουμε να γίνει μια λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτό που ονομάζουμε αναθεώρηση των αποτελεσμάτων, κάτι που θα μας επιτρέψει να αναλύσουμε τα προγράμματα με γνώμονα όλους τους στόχους. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουμε παραχωρήσεις όσον αφορά τη διατήρηση φιλόδοξων στόχων που ορίστηκαν στα προγράμματα για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο. Επίσης θα προσπαθήσουμε να κοινοποιήσουμε, να, να επικοινωνήσουμε αυτό που κάνουμε. Όπως ξέρετε πολύ σωστά, βασιζόμαστε στα στοιχεία που μας δίνουν τα κράτη-μέλη, στις διάφορες πληροφορίες που μας παρέχουν και χαίρομαι που βλέπω ότι σύμφωνα με το ελεκτικό συνέδριο το 95% των αποτελεσμάτων αυτών ε, θεωρούνται αξιόπιστα. θα ήταν μεγάλη δυναμία να μην, του συστήματο διαχείριση και ελέγχου να μπορούμε να βασιστούμε στα στοιχεία των κρατών μελών. Αυτό θα δημιουργούσε αυτόματα πάγωμα ή αναστολή των πληρωμών, έτσι όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Σε κάθε περίπτωση διαπιστώνουμε ότι οι εθνικές αρχές προσέχουν πολύ περισσότερο όσον αφορά την περίοδο σε σχέση με την περίοδο 7 έως 14 όσον αφορά τη διαδικασία διαβίβαση δεδομένων. Γιατί, διότι γνωρίζουν ότι ε, είναι αρκετά μεγάλες οι απειλές. Ε, είχαμε μία έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου όπου οι αρχές έλεγξαν τα αποτελέσματα βάσει κάποιων ελεκτικών διαδικασιών όπως είχαν προβλεφθεί από τους κανονισμούς. Ωστόσο, το θέμα που εξετάζουμε εδώ είναι πολύ σημαντικό και περίπλοκο με όλα τα προβλήματα που αναφέρατε. Αυτό μάλιστα σχετίζεται και με θέματα εμπιστοσύνη στι εθνικές ελεγκτικέ αρχές για μένα είναι βασικότατο αυτό το πρόβλημα. Χρειάζεται να μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στις εθνικές ελεγκτικέ αρχές. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι είναι ανεξάρτητε και ότι λειτουργούν ανεξάρτητα και ότι οι πολίτε. Ε, θα είναι βέβαιοι ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρησιμοποιούνται για τον απότερο στόχο για τον οποίο έχουν προοριστεί, δηλαδή τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Γι' αυτό το λόγο με το ελεγκτικό συνέδριο προσπαθούμε να υλοποιήσουμε αυτή την αρχή του μοναδικού ελέγχου, του ενιαίου ελέγχου. Πρέπει να προσέχουμε να μην έχουμε επικαλύψεις. Ε, το θέμα είναι να αλληλοσυμπληρωνόμαστε πρέπει να μπορούμε να βασιστούμε στη δουλειά των εθνικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να μπορούμε και να συνεχίσουμε και να αξιοποιούμε σωστά τους ελεκτικούς μας πόρους που όπως σας είπα είναι περιορισμένοι. Ε, επικεντρωνόμαστε λοιπόν και βασιζόμαστε και στη δουλειά των εθνικών αρχών ε, και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους κινδύνους. πριν πούμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στις ελεγκτικές αρχές πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες διασφαλίσεις όσον αφορά την ποιότητα της εργασίας των αρχών αυτών. Εξέτασουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν, τις διαδικασίες που εφαρμόζουν και μετά κάνουμε νέο έλεγχο ε, για τι δραστηριότητε που λαμβάνουν χώρα τόπου ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε κατά πόσο το ποσοστά ασφάλματο που αναφέρονται αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Θέλουμε να ξέρουμε ότι μπορούμε να υπολογίζουμε στις ε, ελεγκτικές αρχές λοιπόν και στο έργο τους και στο ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν τέτοιε ε, τέτοιες ποιότητες εργασίας, εργασία. Όπως ξέρετε στην προγραμματική περίοδο η Κομισιόν θεωρήσε ότι πάνω από 330 ελεγκτικές ε, δραστηριότητες είχαν επιτελέσει το, το έργο αλλά δεν εφησυχαζόμαστε. Ε, θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την εργασία των ελεγκτικών αυτών αρχών με στόχο να αποφευθούν κενά και ελλείψεις στο μέλλον. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται με την παραγωγή σωστών αποτελεσμάτων. Όπως είπα πέρυσι, προσπαθήσαμε να αποφύγουμε ε, την επανάληψη των ίδιων ελέγχων με το ελεγκτικό συνέδριο Κάναμε ελάχιστου ελέγχου στα προγράμματα, διότι δεν είχαμε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων που να πετούν τέτοιο έλεγχο. Για φέτος ε, έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν προγραμματωστεί 58 έλεγχοι, 19 αποστολές επιτόπου, ώστε να επιληθευτεί η δουλειά των ε, ε, ελεγκτικών αρχών όσον αφορά τον προσδιορισμό των κινδύνων, την ανείχνευση των κινδύνων και αυτό θα μας επιτρέψει του χρόνου στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων να πούμε αν ε, ε, τα ποσοστά ασφάλματος ε, και οι έλεγχοι των κρατών μελών αντιστοιχούν ή όχι στην πραγματικότητα ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν σημειώνονται σημαντικά ελλείμματα. Όπως είπα, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε να παρέχουμε βοήθεια στις ελεγκτικές αρχές ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι εργάζονται σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες. Και στο ίδιο επίπεδο, διότι σε ορισμένες χώρες διαπιστώσαμε ότι οι ελεγκτικές αρχές και οι διαχειριστικές αρχές ήταν δύσκολο να τηρήσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εμείς παρήχαμε τη σχετική βοήθεια όσον αφορά τα προβλήματα με τα οποία είχαν να κάνουν οι διάφορες αρχές, κυρίως όσον αφορά τις μεθόδους, τη δειγματοληψία, την επεξεργασία των δεδομένων, την προσέγγιση ανάλογα με τον τομέα, τα χρηματοδοτικά μέσα και άλλα στοιχεία όπως είπατε και εσείς. Ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, δυστυχώς, το πρόγραμμα που είχαμε μας επέτρεψε να μείνουμε στο επίπεδο σημαντικότητας του 2%. Ξέρετε ότι είναι προσωρινό το πρόγραμμα που έχουμε στον ιστορικό κανονισμό. Μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε ελέγχου όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, και όσον, αλλά όχι όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Τράπεζα Επενδύσεων. Οπότε οι ελεκτικέ αρχέ ε, των χωρών όπου υπήρξε το πρόβλημα δεν είχαν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν ελέγχου. Μετά άλλαξε ο κανονισμό μέσω του Omnibus. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν το ελεκτικό συνέδριο εντόπισε τις ελλείψεις, τα προβλήματα επιλύθηκαν, αλλά οι συντελεστές σφάλματος παρέμειναν ε, Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν. Να σα πω λοιπόν πω δεν μπορούμε να ξεχνάμε εδώ τη σημασία που έχουν τα χρηματοπιστικά μέσα συνολικά. Γιατί όπω σα είπα, είχαμε μία υπόθεση σε ένα κράτο μέλο ένα πρόβλημα μεγάλης κλίμακος και κατά τη γνώμη μας η εφαρμογή των χρηματοπιστικών ε, ε, μέσων ε, σε αυτή την περίπτωση με δημοσιονομικούς περιορισμούς είναι ο καλύτερος τρόπος για να παγιώσουμε τον αντίκτυπο που έχουν τα δικά μας προγράμματα και γι' αυτό θα σας ζητούσα το ποσοστό επιλογής για την προγραμματική περίοδο να θεωρήσετε πως βρίσκεται στο 74,4% τουλάχιστον αν όσον αφορά τα ταμεία συνοχής, όπως επίσης και το, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Να σας πω πως το ποσοστό εφαρμογής για τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία ε, είναι πολύ ενθαρρυντικά. Έχουμε κάνει μεγάλα βήματα και θα καταφέρουμε να πλησιάσουμε τους στόχους που είχαμε βάλει στα πλαίσια ε, του ε, Ευρωπαϊκού Επενδυτικού προγράμματος. Είχαμε μια αύξηση της τάξης του 95% και πρέπει να σας πω πως για την ε, χρηματοδότηση μέσω χρηματοδοτικών εργολείων αυτό σημαίνει πως τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να πληρώσουν τους ε, τελικούς αποδέκτες πριν λάβουν τη δεύτερη δόση της ε, χρηματοδότησης. Τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος ε, ο και βασικότερος λόγος για τον οποίο έχουμε αυξημένα ποσοστά σφάλματος. Και να σας πω πώς ξεκινήσαμε πρώτα απ' όλα με δημόσιες, με κρατικές προμήθειες. Γιατί ξέρετε πως στους κλάδους αυτούς έχουμε τα περισσότερα σφάλματα. Τώρα, περνάμε και σε μία ε, φάση που τα ποσοστά εκεί είναι πραγματικά χαμηλά και τα σφάλματα τα βρίσκουμε τώρα πιο πολύ εκεί που υπάρχουν χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Και το ζήτημα εδώ ε, που αυξάνει το ποσοστό σφάλματος είναι το αποδεκτό ε, αυτών των ε, προγραμμάτων, δηλαδή το κατά πόσο θα έπρεπε να έχουν εγκριθεί ή όχι. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ υπέρ του να βρεθούν οι λόγοι ε, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα κυνήγι μαγισσών γιατί δεν είναι πρόβλημα αφορά η Νότου ή κάποια συγκεκριμένη χώρα. Είναι ακριβώς όπως το είπατε εσείς. Και το είπε και η Πρόεδρος με την περίπτωση της Τσεχίας. Τα προβλήματα δεν είναι προβλήματα των Ταμείων Συνοχής ή του ΕΤΠΑ τα προβλήματα αυτά κάποτε ναι σχετιζόντουσαν με τα δικά μας ταμεία και με το γεγονός πως οι αρχές ε, ενέκριναν και μετά α, απεντάσανε προγράμματα και έργα τα οποία είχαν χρηματοδοτηθεί με δικά μας ταμεία και τελικά σε, όταν φτάναμε στην τελική ε, πληρωμή είχαμε πρόβλημα. Αλλά κάνοντας με μία συμφωνία που κάναμε με την Όλαφ, με την οποία συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά, και από την οποία λαμβάνουμε εκθέσεις σχετικά με τα δικά μας ταμεία, πρέπει να σας πω πως μας έστειλαν κάποιες συστάσεις τις οποίες εμείς εφαρμόσαμε κατά γράμμα. Έτσι λοιπόν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περιοχή της Βοημίας, κεντρικής Βοημίας ή για τα περιφερειακά ταμεία ε, να σας πω πως η τσεχική κυβέρνηση ζήτησε αυτά τα αιτήματα χρηματοδότησης να αποσυρθούν και πια δεν έχουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Το πρόγραμμα έκλεισε. Χωρίς αυτά. Τώρα για την κατάσταση. Της Eurofair που συζητήθηκε και από την Τσεχική Βουλή, να σας πω πως λόγω ακριβώς του οικονομικού κανονισμού που έχουμε, θεωρήθηκε πως είναι ευθύνη των εθνικών αρχών. Η λήψη μέτρων για να προλαμβάνεται η σύγκρουση συμφερόντων είναι θέμα εθνικής νομοθεσίας. Και αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα των εθνικών αρχών. Ακριβώς γιατί πρόκειται για δαπάνες που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό και ακολουθώντας την αρχή της πολυμερούς διαχείρισης οι αρχές, ε, οι εθνικές, θα πρέπει να αναλάβουν στο σημείο αυτό τις ευθύνες τους. Γι' αυτό ζήτησα πληροφορίες επιπλέον για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι ώστε να καταφέρουμε να αξιολογήσουμε πραγματικά πώς έχει η κατάσταση. Είπατε κι εσείς πολύ σωστά πως τα στοιχεία που μας έστειλε η Διεθνής Διαφάνεια για το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων ε, κυρίως το πρόβλημα είναι με αυτό τον όμιλο, την Αγκροφέρ και οι αρχές μας έστειλε κάποιες πληροφορίες για τα τόσο συμβαίνουν στην Δημοκρατία της Τσεχίας αυτό κατόπιν αιτήματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τις πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνουμε πως πολλές εταιρείε οι οποίες συνδέονται με την Αγκροφέρτ έλαβαν επιδοτήσεις και ενισχύσεις έτσι και μετά για το λόγο αυτό προχωρήσαμε εμείς σε ανακτήσεις και σε απόσυρση ε, των ε, ε, χρηματοδοτήσεών μας. Αύριο νομίζω ο κύριος Χόγκαν θα μπορέσει να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες ε, για τα θέματα με τα γεωργικά ταμεία. αλλά για τα ταμεία τα οποία διαχειριζόμαστε εμείς, που είναι αυτά της περιφερειακής ανάπτυξης, και τα περιφερειακά ταμεία δεν έχω κάτι παραπάνω από τώρα για το θέμα της Ουγγαρίας. Να σας πω λοιπόν. Η Ουγγαρία εξέφρασε ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο ε, ανατέθηκαν κάποιες συμβάσεις και οι δικές μας υπηρεσίες ενημέρωσαν και πέρσι και φέτος μας ενημέρωσαν πως στην Ουγγαρία παρακολουθούμε στενά το θέμα της ανάθεσης ε, κάποιων συμβάσεων σε περίπτωση που υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για τις κρατικές προμήθειες και κοιτάμε το πώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια από τα Ταμεία Συνοχής και πιο συγκεκριμένα να σας πω πώς στην περίπτωση στην οποία έχει επέμβει η Όλαφ ζητήσαμε από τις Ουγγρικές Αρχές να μας δώσουν περισσότερες προφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση αυτών των ε, κρατικών προμηθειών. Εν πάση περιπτώσει παροτρύνουμε αυτό το κράτος μέλος να υποστηρίξει τον θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων τουλάχιστον ε, στην περίπτωση των ε, ε, κρατικών συμβάσεων και των αναθέσεων στις κρατικές προμήθειες. Αυτή τη στιγμή οι ουγγρικές αρχές διαφωνούν με τα αποτελέσματα που έχουμε εμείς διαπιστώσει. Οπότε, κάναμε μια καινούρια μελέτη σε 10 κράτη-μέλη ένα από αυτά είναι η Ουγγαρία για να δούμε τι γίνεται με τη διαδικασία ε, απευθείας ανάθεσης και για τα ερωτηματικά αυτά τα οποία προκύπτουν όταν, για παράδειγμα, ε, όταν είναι μία και μοναδική εταιρεία η οποία κατεβαίνει σε ένα διαγωνισμό με υψηλό προϋπολογισμό. Ελπίζω πως θα λάβουμε περισσότερες πληροφορίες και θα σας ενημερώσουμε. Ε, Πολλά κράτη-μέλη, και εδώ θα συμπεριλάβουμε και την ε, Τσεχία και την Ουγγαρία, ε, αντιμετωπίζουν ε, τέτοιου είδους κινδύνους όταν έχουμε διαγωνισμούς, όταν έχουμε κρατικές προμήθειες και αναθέσεις. Παρακολουθούμε το θέμα αυτό στενά και εμείς έχουμε στόχο να προτείνουμε συγκεκριμένες διαδικασίες στα πλαίσια της ελεγκτικής διαδικασίας. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, για τις πληρωμές. Δυστυχώς η Ουγγαρία είναι πολύ ψηλά στον κατάλογο αυτών που έχουν ε, δημοσιονομικές διορθώσεις μιλάμε για δισεκατομμύρια και να σας πω πως σχετικά με τα κράτη-μέλη εμείς αυτό που βλέπουμε είναι πως ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν επηρεάζεται. Γιατί, Γιατί εμείς επιβάλλουμε στο 100% τις διορθώσεις όταν μας το ζητά η Όλαφ. Και τα κράτη-μέλη και οι κυβερνήσεις τους καλό θα είναι να απευθυνθούν μετά στις ε, εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για να επιστραφούν ε, τα ε, αχρηστήτως αυτά κατεβληθήντας στον εθνικό προϋπολογισμό. Νομίζω δεν άφησα τίποτα έξω. Και άλλη ερώτηση. Και... Τρεις, τρεις συνάδελφοι θέλουν να ρωτήσουν. Ο συνάδελφος Φόρς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για τις απαντήσεις που στείλατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά Δεδομένου ότι υπήρξε αυτή η έκθεση για την τσεχική δημοκρατία, υποχρεωμένα να παρέμβω. Το ζήτημα αφορά αυτή την καταγγελία της Transparency International, της Διεθνούς Διαφάνειας. Καταγγελία η οποία θα ακολουθήσει την τυπική διαδικασία. Η υπόθεση αυτή του Αντρέ Μπάμπης είχε και διάφορες εξελίξεις τις τελευταίες εβδομάδες. Χρειαζόμαστε λοιπόν την ακριβή άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά αυτό το ζήτημα σύγκρουση συμφερόντων και κατά πόσο αυτές οι, κρατικές, ε, οι οικονομικές ενισχύσεις ε, αποτελούν κατάχρηση. Πρέπει να ξέρουμε πώς έχουν ακριβώς τα πράγματα με τον Άντρε Μπάμπης, διότι πλέον δεν διαχειρίζεται αυτή την επιχείρηση, δεν διευθύνει πλέον αυτή την επιχείρηση, αφού η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ψηφίσει αυστηρότατη νομοθεσία όσον αφορά τις σύγκρουση συμφερόντων. Τις ε, χρειαζόμαστε όλες αυτές τις πληροφορίες, ε, θεωρώ. Και επίση πρέπει να μάθουμε τι πορεία έχει ακολουθήσει αυτή η καταγγελία και τι έχει γίνει με αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Με ποιο τρόπο λοιπόν η Κομισιόν πρόκειται να μας ενημερώσει για το αποτέλεσμα της διαδικασίας και για την καταγγελία της Transparency International θα πάρει εβδομάδες, μήνες. Ίσως να μην έχετε ακόμα απάντησης για αυτές τις ερωτήσεις, αλλά όταν θα έχετε μπορείτε να μας τις στείλετε γραπτός. Αύριο στις 12 θα συνεδριάσουμε με τη Γενική Διεύθυνση Αγκράρ και θα συζητήσουμε ακριβώς αυτά τα θέματα. Η συνάδελφος Ρέντα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Είναι σαφές ότι το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων του Πρωθυπουργού Μπάμπης είναι πολύ σημαντικό για τα μέλη. Κυρία Επίτροπε, πρέπει να πω ότι δεν σύμφωνο με την ερμηνεία ότι η πρόληψη της σύγκρουσης είναι 100% ευθύνη κρατών μελών. Ο δημοσιονομικός κανονισμός λέει ότι αυτή η υποχρέωση περιλαμβάνει τις εθνικές αρχές, αλλά δεν περιορίζεται που δεν είναι σε αυτές. Αφορά ονδήποτε εμπλεκόμενος στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ή τον έλεγχο. Ε, η ερμηνεία η δικιά μου είναι ότι σαφώς περιλαμβάνει, ε, περιλαμβάνεται εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τονίζω γι' αυτό το λόγο ότι βέβαια αν το κόμμα των πειρατών και η διεθνής διαφάνεια ασχολη, ε, αναφέρθηκαν στην Κομισιόν για αυτό το θέμα, αυτό έγινε συγκεκριμένα γιατί δεν περίμεναν πολύ βοήθεια από τις εθνικές αρχές τους, ε, ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ύποπτος και ο ανακρινόμενος είναι ο Πρωθυπουργό. Και σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του κυρίου Μπάμπη ε, ω το ελεγκτή του Αγκρόπαρτ, έπρεπε να πάνε στη Σλοβακία για να βρουν τις πληροφορίες που δεν υπήρχαν στη τσεχική δημοκρατία και δεν τι έδιναν οι τσεχικές αρχές. Ρωτώ λοιπόν θα γίνει... Ε, α, ε, έγινε μια συνάντηση με τον κύριο Μπάμπη στις 6 Σεπτεμβρίου, έτσι μαθαίνω, όπου στη συζήτηση αυτή είπατε και για το θέμα των επιδοτήσεων κύριο, στην εταιρεία AgroFed του κυρίου Μπάμπης και συζητήσατε και για την εκτέλεση της πολιτικής συνοχής στην Τσεχία και την πρόταση της Κομισιόν για την επόμενη πολιτική συνοχής. Και επειδή η Κομισιόν έχει υποχρέωση βάσει του άρθρου 61 του δημοσιονομικού κανονισμού να προλαμβάνει τη σύγκρουση συμφέροντων, αλλά και να ασχολείται με οποιοδήποτε τυχόν τέτοιο πρόβλημα. Τι δράση αναλάβατε κατά τη συνάντηση με τον κύριο Μπάμπης ώστε να λυθούν τα κατάλληλα μέτρα. Δεύτερον, λαμβάνοντα υπόψη ότι το κόμμα των πειρατών διαπίστωσε ότι ο κύριος ε, Μπάμπης ε, ε, ήταν και ο δικαιούχο και ο πάροχος, σε τελευταία ανάλυση ο κύριος Μπάμπη ελέγχει την Αγροφέντ σε, σύμφωνα με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με εφορίας. Βλέπετε εσείς κάποια δυνατότητα παρά το γεγονός ότι έγινε σαφής αναφορά ότι ο έλεγχος περιλαμβάνει και την εταιρεία και τον δικαιούχο. Μπορεί ο κύριος Μπάμπης να μην είναι ο ελεγκτής της συγκεκριμένης εταιρείας Agrofed. Και ο τελευταίος ομιλητής μας. Έχω. Α.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 Αξιότιμε επίτροπε, είναι μεγάλη μου χαρά που όποτε σας ορίζω για να μιλήσουμε για την πολιτική συνοχής και τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Τώρα, για το γενικό προϋπολογισμό ήδη μιλήσαμε διεξοδικά και πώς μπορούν να εκπροσωπηθούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Είναι εδώ σημαντικό να εντοπίσουμε τα κακό κείμενα σε σχέση με τα ταμεία. Συγκεκριμένο παράδειγμα από την Ουγγαρία που δείχνει ότι δεν αρκεί να επισημαίνουμε τα κακό κείμενα αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε και στις νομικές επιπτώσεις. Η εταιρεία Ήλιο στην Ουγγαρία είναι μια επιχείρηση η οποία κάποια στιγμή κέρδισε 13,5 δις μέσα από διαγωνισμούς της Ένωσης. Και η εταιρεία αυτή, η οποία συνδέεται με τον Πρωθυπουργό, όπως φάνηκε, ε, δεν ε, λειτουργούσε σωστά. Δηλαδή σε συγκεκριμένες περιόδους και σε σχέση με συγκεκριμένες διασυνδέσεις ε, δεν ήταν εντάξει. Και έτσι ζημιώθηκαν και τα συμφέροντα της Ένωσης. Άρχισε λοιπόν μία έρευνα η οποία Ε, ε, ε, τερματίστηκε γιατί δεν εντοπίστηκε αδίκημα. Τη στιγμή που θα έπρεπε να προχωρήσει η Όλαφ, γιατί υπήρχαν αποχρώσεις ενδείξεις, ε, έπαυσε η διαδικασία, είπαν ότι δεν υπάρχει ε, αδίκημα. Και αυτό είναι συνέπεια, δείχνει ασυνέπεια. Και βλέπετε πώς είναι, ε, ότι υπάρχει ανάγκη ανάληψη δράση της Ένωσης και της Κομισιόν συγκεκριμένα. Η Όλαφ κατέδειξε κάποιο πρόβλημα, ενώ υπονομεύτηκε η περαιτέρω διαδικασία από το, τη συγκεκριμένη χώρα μέλος. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν συγκεκριμένα, ούτως ώστε να συναχθούν ε, τα απαραίτητα συμπεράσματα να κατησχύσει ο νόμος και να προστατευτούν οι, κατα... οι φορολογούμενοι. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί όταν αυτοί οι ε, λογαριασμοί αποκλειστούν από τους λογαριασμούς που αποστέλλονται και τις απαιτήσει που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, θα υπάρξει λογοδοσία. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Μέχρι πότε θα ανέχεται η Κομισιόν να αποστέλουν λογαριασμούς τα κράτη-μέλη που δείχνουν ότι εδώ υπάρχει διαφθορά, υπάρχουν καταχρήσεις. Και παρόλα αυτά συνεχίζουν και πολλές φορές απλώς αποσύρουν την αξίωση και δεν υφίστανται καμία κύρωση. Αυτό δεν είναι καλό για την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια και τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης δεν διαφυλάσσονται, ούτε καταπολεμείται η διαφθορά. Και για μετά το 2020 θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε να βρούμε απλούς και, αλλά και αποτελεσματικούς τρόπους για να υπάρχει λογοδοσία και να ισχύει ο νόμος, να, αντιμετωπίζουν τις νομικές επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζέντερ, κυρία Επίτροπε. Και εγώ σας καλωσορίζω όπως οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση και μια ερώτηση παρακαλώ πολύ. Η παρατήρησή μου είναι η εξής. Από ό,τι γνωρίζω, και αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε κάποια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι εξουσιοδοτημένη ε, για να ερευνά τον Πρωθυπουργό της Τσεχίας. Οι νομικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διατάξεις των κρατών μελών προβλέπουν ότι η Τσεχική Δημοκρατία είναι ένα κράτος μέλος ε, μετά από ελεύθερες εκλογές όπου οι Τσέχοι πολίτες έριξαν την ψήφο τους και το κόμμα που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους ε, διόρισε τον Πρωθυπουργό που εκλέγεται από το Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η διαδικασία. Η ερώτηση τώρα είναι, η κυρία Επίτροπος θα δει ε, ε, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το βρίσκει σωστό ότι ο πρόεδρος Μακρόν η ε, ε, ε, συμπαθεί την Γερμανίδα Καγκελάριο ή όχι, γιατί από ό,τι ξέρω εγώ τα πολιτικά γούστα και οι προτιμήσεις δεν έπαιξαν ποτέ ρόλο ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ερώτησή μου τώρα. Μπορεί να πει κανείς ότι η Όλαφ δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Και αυτό δημιουργεί δυσκολίες και για το Κοινοβούλιο και για την Κομισιόν. Υπάρχουν δύο στοιχεία που αποδεικνύουν, θα έλεγα, ότι η Όλαφ δεν εργάστηκε καλά. Εγώ δεν θα πω τώρα αν υπάρχουν πολιτικές διασυνδέσεις, ε, ότι, ε, που, που ε, ότι δηλαδή ο επικεφαλής της Όλαφ είναι ένας ε, παλιός αριστερός και ότι οι έρευνες γίνονται σε μια εποχή όπου ε, επίκυνται εκλογέ στην Τσεχία. Και έτσι κι αλλιώς ο, ο άνθρωπος για τον οποίο μιλώ δεν είναι πια στην Όλαφ. Τώρα το ένα είναι η καρδιά της Βουδαπέστης και το άλλο είναι το πρόγραμμα Ήλιος. Η Όλαφ έκανε πολύ συγκεκριμένες διαπιστώσεις. Στη μία περίπτωση η Γενική Διεύθυνση της, της Κομισιόν δεν ήταν σύμφωνη με τις διαδικασίες της Όλαφ και ούτε συμφώνησε με τις διαπιστώσεις της Όλαφ και είπε ότι δεν συντρέχουν ε, λόγοι για έρευνα και δεν υπάρχουν κακοσκίμενα Και στην περίπτωση του Ήλιος, οι ουγγρικές αρχές διεξήγαγαν τις έρευνες και πάλι κατεδείχθη ότι η Όλαφ δεν εργάστηκε σωστά που είχε διαπιστώσει, δηλαδή η Όλαφ ότι εδώ πρόκειται για κάποιο αδίκημα. Όχι, η Γενική Διεύθυνση δεν επιβεβαίωσε κάτι τέτοιο. και δεν πρέπει να έρχονται οι γενικές διευθύνσεις και οι επίτροποι σε άσχημη θέση διότι η Όλαφ ε, έκανε κακής ποιότητας δουλειά και τα στοιχεία που έδωσε δεν είναι σωστά. Δεν ε, τεκμηρίωσαν ενδείξεις για συνέχιση της έρευνας. Δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Η ερώτηση είναι λοιπόν, δεν ήρθε η ώρα να ανακαλέσουμε σε κάποια τάξη την Όλαφ, ούτω ώστε η τελευταία να μην εργάζεται ε, ως ε, ε, αρχή ε, υπεράνω όλων των διατάξεων. Η έρευνα ήταν εξαιτία εξαιρετική, η αυτά ήταν εξαιρετική στην Όλαφ. Ε, υπήρχαν κάποια θέματα σε σχέση με τη καρδιά της Βουδαπέστης. Ε, ούτε πρόκειται για προτιμήσεις ή γιγούστα, ούτε πρόκειται για επίκριση της εκλογικής διαδικασίας. Ε, το θέμα είναι ότι η επικεφαλής ο αρχηγός, ο πρόεδρος της κυβέρνησης δημιούργησε πρόβλημα ε, που ερμηνεύεται ως σύγκρουση των συμφερόντων. Ε, ενδεχομένως ε, και γι' αυτό η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών έπρεπε να κάνει κάποιες ερωτήσεις. Η κυρία Επίτροπος έχει το λόγο. Κυρία Κρέτσου. Ευχαριστώ πολύ. Τι κρίμα, τι κρίμα που το θέμα αυτό έχει πολιτικοποιηθεί τόσο πολύ. Γιατί εδώ Μιλάμε για συγκεκριμένες υποθέσεις και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να περιοριζόμαστε σε κάτι τέτοιο. Ε, τουλάχιστον όχι για την περίπτωση της ε, δημοκρατίας της Τσεχίας. Και να σας πω πως εγώ είμαι επίτροπος για την περιφερειακή ανάπτυξη και πιστεύω πως η εφαρμογή και η εκτέλεση προχωρά σωστά. Δίνει καλά αποτελέσματα, τουλάχιστον σε επίπεδο ε, Ταμείων Περιφερειακής Ανάπτυξης και στα Ταμεία της Συνοχής. Τώρα, για τις πρώτες πληρωμές που έγιναν, νομίζω ότι πάμε καλά. Για την Τσεχία τώρα και την Ουγγαρία, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιορίζουμε την εικόνα που βλέπουμε σε αυτές τις συγκεκριμένες υποθέσεις τις οποίες εδώ θίξαμε. Και θα ήθελα να δώσω μία απάντηση στον κύριο Ντόιτς. Εγώ σέβομαι απόλυτα όλους τους προέδρους, όλους τους πρωθυπουργούς που έχουν εκλεγεί από τα κράτη-μέλη. Στις 6 Σεπτεμβρίου πήγα στην Τσεχία. Είναι μια χώρα σημαντική. Και πρέπει να σου πω πως συναντήθηκα με τον πρωθυπουργό, όχι με πρόεδρο επιχείρησης Διοικητικό Σύμβουλο και μάλιστα πρέπει να σας πω πως δεν πήγα μόνη μου, πήγα με τους συναδέλφους από την DG Regio για να μιλήσουμε για την ανάγκη επιτάχυνσης της εκτέλεσης των προγραμμάτων και για το κρίσιμο σημείο από εμά είναι μια συμφωνία στα πλαίσια ε, του Συμβουλίου το επόμενο έτος που θα γίνει υπό Ρουμανική ε, Προεδρία στο CBU γιατί εκεί θα πρέπει να δούμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, να το συμφωνήσουμε, έτσι ώστε να μην έχουμε άλλες καθυστερήσεις για όλη την περίοδο εκτέλεσης ε, εκείνη. Η απάντηση που έλαβα ήταν πάρα πολύ δεκτική, πολύ ανοιχτή στις ερωτήσεις που έκανα. Μίλησα και με εκπροσώπους ε, των διαφορών κομμάτων και με το κόμμα των πειρατών. αξιολογήσαμε την κατάσταση και είπαμε ότι μέχρι τον Ιανουάριο θα δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήσεις που μας έκαναν ε, στην Τσεχική Βουλή. Δυστυχώς δεν έχω ακόμα περισσότερες πληροφορίες για να σας μεταφέρω για τη συνάντηση αυτή. Αυτά που μας είπε ο πρόεδρος ή η πρόεδρος σας ε, δεν έχω κάτι να προσθέσω παραπάνω. Όμως, θα ήθελα να πω το εξής. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, εδώ η κατάσταση είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Και εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μία γνωμοδότηση πριν λάβουν το λόγο πιο επίσημοι θεσμοί, γιατί δεν θέλουμε να πολιτικοποιηθεί η υπόθεση. Για την περίπτωση και την υπόθεση στην Ουγγαρία, εκεί τρέχει αυτή τη στιγμή μία έρευνα. Ξέρετε και εσείς οι Ουγγρικές αρχές δεν συμφωνούν με τα όσα έχουμε εμείς πει, τουλάχιστον για το πρόγραμμα Ήλιος. Εκεί τα πράγματα δεν ε, έχουν κλείσει και δεν θα κλείσουν μέχρι να πιστούμε μέχρι να λάβουμε τα τελικά συμπεράσματα της Όλαφ για το κατά πόσο είναι ε, απαραίτητο να επιβάλλουμε οικονομικές κυρώσεις ή όχι. Θα ήθελα επίση να πω το εξή. Για την ε, περίοδο 14-20 εμείς συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις Ουγγρικές Αρχές για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τους κινδύνους σχετικά με τις κρατικές ε, ε, προμήθειες, όπως επίσης και με την επιλογή των έργων. Όπως ε, σας είπα, πρόκειται να γίνει μια προληπτική αποστολή αξιολόγησης σε διάφορα κρατημέλη, ένα από αυτά είναι η Ουγγαρία, και μετά θα είμαι καλύτερα προετοιμασμένη για να μπορώ να απαντήσω στις δικές σας ερωτήσεις. Όμως, θα πρέπει να πω το εξής. Ας περιοριστούμε σε αυτά τα δύο κράτη, γιατί γενικά μιλάμε για το θέμα της απάτης. Και προσωπικά πιστεύω πως τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά και έχουμε αποδείξει πως έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία κάθε χρόνο και πως έχουμε δώσει ευκαιρίες να εντοπίσουμε την απάτη που γίνεται με ευρωπαϊκά κονδύλια. Η απάτη αυτή τη στιγμή είναι το 0,4% για την πολιτική συνοχής. Και θα το επαναλάβω για μια φορά ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πεπισμένη πως θα αντιμετωπίσει με στεναρότητα τις περιπτώσεις διαφθοράς και απάτης. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοιχτούμε κάτι τέτοιο. Έχουμε λάβει πολύ σημαντικά μέτρα για τα θέματα αυτά και για την περίοδο 14-20 για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να πατάξουν τη διαφθορά και την απάτη. Και αυτή είναι και η υποχρέωσή μας, νομικά ομιλώντας, να δώσουμε τη μάχη κατά της απάτης Και να σας πω πως για τις εθνικές αρχές ελέγχου έχουν ληφθεί μία σειρά μέτρα και δυστυχώς μέχρι στιγμής ε, δεν ήταν υποχρεωτικά αυτά, αλλά πολλά κράτη-μέλη σε θελοντική βάση αποφάσισαν πως ο καλύτερος τρόπος είναι να ενισχύσουμε τη δράση, να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή απόκριση, έτσι ώστε αυτές οι παραβιάσεις να μην λαμβάνουν χώρα. Πολλοί θα βρεθούν λοιπόν ενώπιον των δικαστηρίων και αυτό θα έχει και αποτρεπτικό ρόλο. Και εσείς μάλιστα πρέπει να σας πω ξεκινήσατε την όλη διαδικασία για να διορίσετε ε, αυτό το γενικό εισαγγελέα που θα αναλάβει το θέμα αυτό. Τώρα, να σας πω πως αυτές οι παρατυπίες καμιά φορά δεν είναι απάτη. Για παράδειγμα, στις διαγωνισμούς κάποιες διαγωνιστικές διαδικασίες δεν γίνονται με τον καλύτερο τρόπο ή δεν γίνονται σεβαστές. Και για να εντοπίσουμε όλα αυτά χρειάζεται μια πολύ στενή συνεργασία με την Όλαφ. Έτσι μόνο θα πατάξουμε την απάτη σε όλα τα ταμεία και στα ταμεία συνοχής και πρέπει να σας πω πως στόχος μας είναι σε συγκεκριμένους κλάδους να ενισχύσουμε τη συνεργασία με την Όλαφ έτσι ώστε να κάνουμε και προληπτικούς ελέγχους οι οποίες θα βασίζονται στις συστάσεις ακριβώς που μας έχει δώσει η Όλαφ. Αυτό είναι μια πάθωση που έχουμε πάρει συλλογικά και είμαστε ικανοποιημένοι γιατί στο παρελθόν δεν είχαμε ποτέ αυτό το επίπεδο συνεργασίας, δεν είχαμε ποτέ τέτοιες υποθέσεις ε, σχετικές με τα ευρωπαϊκά κονδύλια όπου ένα τόσο υψηλό κομμάτι ε, του προϋπολογισμού μας να εμπλέκεται. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την διαδικασία πλούστευσης και είμαι στη διάθεσή σας εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις ή αν θέλετε να σας κάνω κάποια περαιτέρω ενημέρωση. Ich fürchte, wir sind jetzt fast am Ende unserer zeitlichen Möglichkeiten. Das Wort erhält noch Herr Murphy vom Rechnungshof. Bitte auch noch mit einem Hin. Ήθελα να δώσω στο, το λόγο στο ελεκτικό συνέδριο για να μας παρουσιάσει τη νέα μεθοδολογία και μετά στην ε, εισηγήτρια. Έχετε το λόγο, το ελεγκτικό συνέδριο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όπως είπαμε και στην παρουσίαση υπάρχει μια συγκεκριμένη προσέγγιση. Όπως είπε η Κομισιόν, είναι καλό που έχει μειωθεί το ποσοστό σφάλματος. Όπως είπαμε, το 1% ήταν από ένα χρηματοδοτικό μέσο μόνο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε όπως είπαμε, ε, κάποιες από τις σημαντικές προκλήσεις για το 2017 ήταν ότι είχαμε κοιτάξει περιορισμένες δαπάνες και λίγες αρχές και δεδομένων των ελλείψεων που διαπιστώσαμε υπάρχει περιθώριο για βελτίωση ώστε να προχωρήσουμε την προσέγγιση. Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα το 2018 πιστεύω γιατί το δείγμα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και οι δαπάνε θα είναι πολύ περισσότερε. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα τη εργασία των αναρχών σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το γενικό μου συμπέρασμα. Και θα ήθελα να προσθέσω, ξέρω ότι έχουμε περάσει τον χρόνο και δυσκολεύεστε λίγο, αλλά όσον αφορά την απορρόφηση, επειδή αναφέρθηκε στην αρχή των συζητήσεων, είναι ένα σημαντικό θέμα. Είδαμε χαμηλά ποσοστά απορρόφηση μέχρι στιγμή 16% νομίζω. Προφανώ, ε, δεν θέλουμε να βλέπουμε απορρόφηση απλά για να υπάρχει απορρόφηση. Θέλουμε σωστή υλοποίηση και επίτευξη των στόχων αλλά βλέπουμε και ένα κίνδυνο. Όταν αφήνουμε τη δαπάνη προς το τέλος του προγράμματος υπάρχει κίνδυνο στα χρήματα αυτά να δαπανηθούν μόνο και μόνο για να δαπανηθούν. Όταν ο πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου παρουσίασε την ετήσια έκθεση στην Επιτροπή Κόντ στο Στρασβούργο, ανέφερε το ποσό των 267 δισεκατομμυρίων. Είναι πάνω από το διπλάσιο από τον ετήσιο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεσμεύτηκε να παρέχει μια αναθεώρηση για να δούμε για ποιο λόγο συσσωρεύονται αυτά τα ποσά και από τις πιο πρόσφατες προφορές που έχουμε ε, η έκθεση αυτή θα κυκλοφορήσει τέλη Μαρτίου. Ευχαριστώ. Η συγγήτρια σύντομα για να τελειώσουμε. Ευχαριστώ και πάλι. Επίτροπε, για τις πληροφορίες και όχι μόνο τις γραπτές. Ευχαριστώ για τη συνεργασία μας και με την ε, Επίτροπε Κρέτσου και με την ομάδα σας. Ευχαριστούμε για τη στενή συνεργασία και τις απαντήσεις σε ερωτήσεις μας. Θέλω να τονίσω κάποια πράγματα. Δηλαδή, εδώ και δεδομένων των εκλογών το 2019 και για να έχουμε τις καλύτερες ε, ε, δυνατότητες διαπραγμάτευσης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και αν πάμε πέρα από την μικροδιαχείριση των απατών ε, που αφορούν συγκεκριμένα ονόματα, πολιτικούς κλπ δούμε το Dieselgate και τη Volkswagen ακόμα δεν ξέρουμε πού είναι οι επιδοτήσεις για να μην μιλήσω και για τη χώρα μου, τη Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε τέτοια. Πρέπει να έχουμε μια θετική προσέγγιση σε όλα αυτά και να είμαστε και ευγνώμονες σε αυτά που λειτουργήσαν καλά, να εντοπίσουμε βέβαια και τα, σε, τους τομείς όπου υπάρχουν προβλήματα αλλά ε, πολλές φορές ε, έχουμε και προβλήματα με υπουργούς και η, η καγκελάριος Μέρκελ ε, είχε το θάρρος να μιλήσει για όλα αυτά και χαίρομαι που κάποιος είχε το θάρρος να πει ότι δεν είναι όλα τέλεια. Ας είμαστε λοιπόν επικοδομητικοί. Ας ενημερώσουμε για τα προβλήματα τους πολίτες μας, ας προσφέρουμε λύσεις με πνεύμα θετικό. Ας εστιάσουμε στις διαδικασίες, ας εστιάσουμε στους κανόνες, στις διαδικασίες μας, ε, να προσπαθήσουμε να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες όσο μπορούμε και να έχουμε περισσότερες, ε, να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη Αυτά τα σκάνδαλα δεν προάγουν την εμπιστοσύνη. Αλλά μην τα ρίχνουμε όλα κάτω από το χαλί, μην τα κρύβουμε. Βέβαια μερικά χαλιά είναι πιο μεγάλα από άλλα. Ας ε, δούμε αυτά τα ανησυχητικά φαινόμενα που μπορούμε να λύσουμε ως Ένωση. Μην δίνουμε την εντύπωση στους ε, πολίτες μας ότι εδώ στο Κοινοβούλιο και, στο, και στην Κομισιόν ε, μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα που πλήττουν την κοινωνία, την κλιματική αλλαγή, τον Ευρωπαϊκό Στρατό, την κλιματική αλλαγή και την καταπολέμηση της ανεργία, της ε, απάτης. Βέβαια ξέρω με τις μεγάλες ε, υποθέσεις απάτης που πολλοί δεν θέλουν να την αντιμετωπίσουν γιατί όλο αυτό είναι μια πολύ δαπανηρή διαδικασία και δεν συνδέεται πάντα με τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Πάντως εμείς θα πρέπει να τους πούμε ειλικρινά στους πολίτες τι μπορούμε να κάνουμε και πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Γιατί στο παρελθόν αυτό που καταφέραμε είναι να βοηθήσουμε τους λαϊκιστές που μας αφαίρεσαν το λόγο. Ε, ευχαριστώ για τη συνεργασία και στο μέλλον είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Νομίζω ότι η ομάδα της κυρίας Κρέτσου θα μας βοηθήσουν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και το ελεγκτικό συνέδριο. Ο κύριος Μέρφυ ήταν πολύ δραστήριος και ευχαριστώ και για τις προτάσεις και για τα σχόλια σας. Να πω ότι δεν έχουμε να κάνουμε με απάτες αλλά με συστημικά προβλήματα, τα οποία συστημικά προβλήματα οδηγούν σε σοβαρή μετατόπιση του ανταγωνισμού μέσα από διαδικασίες της Ένωσης. Δηλαδή εκμεταλλεύονται κάποια παραθυράκια τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Δεν είναι μόνο το θέμα της απάτης. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο καθήκον και προσοχή μην με μεγάλα χαλιά για να κρύβουμε <laughs> πολλά πράγματα από κάτω από αυτά. Αυτό θα ήταν πολύ άσχημο πράγμα. Δεν ε, φαντάζομαι θα συνέβαινε βέβαια κάτι τέτοιο. Ό,τι και να έχει. Ε, να σας ευχαριστήσουμε κυρία Επίτροπε και σας και την ομάδα σας. Θα είμαστε σε επαφή. Δεν το λέω απειλητικά, το λέω φιλικά αυτό. Πάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Ε, πρόκειται για το κλείσιμο των λογαριασμών. Ε, ο κύριος ε, Στάες, ο κύριος Μπαρτ Στάες. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να είμαι σύντομος. Όπως ξέρετε όλοι, η Ολομέλεια στο Στρασβούργο κατά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια απορρίψαμε την απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Αυτό σημαίνει ότι τώρα θα πρέπει να εγκρίνουμε ε, μια πρόταση ψηφίσματος ε, για την πρόταση αυτή για το κλείσιμο των λογαριασμών. Έχουμε υποβάλει μια πρόταση ψηφίσματος. Δεν νομίζω ότι έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Είναι μια διοικητική διατύπωση. Θα πάμε σύμφωνα με τους κανόνες. Λοιπόν, ε, στις 28 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία, στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ. 13 Δεκεμβρίου στην, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και ψήφο στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Τελειώσαμε. Και πάμε στο σημείο 6. Έκθεση πρωτοβουλίας για τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες τη ΕΤΕΠ, τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο κ. Σπυρίνσκι είναι ο εισηγητή και θα μας κάνει την εισαγωγή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την έκθεσή μου. Πώς να το πω, με κάποια ιδιαίτερη δομή όχι κεφάλαιο προς κεφάλαιο. Θα προσπαθήσω να επισημάνω με κάπως αναλυτικό τρόπο τα σημεία που θεωρώ εγώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να λεφθούν υπόψη για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕΠ και του ελέγχου τους. Τι εννοώ πιστεύω ότι πρέπει να επισημάνουμε τρεις βασικές προσδοκίες όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και τον ελεγχό τους. σε σχέση με την ΕΤΕΠ. Πρώτον, πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα της αποστολής που καλείται να επιτελέσει η τράπεζα τόσο δύναμη των συνθήκων ε, όσο και δύναμη του εσωτερικού της καταστατικού. Το να δρά υπέρ της ολοκλήρωσης της ισόρροπης ε, ανάπτυξης ε, και της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Συλλέγοντας από τις κεφαλαγορές σημαντικά ποσά και επενδύοντας τα με ευνοϊκούς όρους ε, σε προγράμματα που προωθούν τους ευρωπαϊκούς στόχους. Δεύτερον, κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία μερικά χρόνια έχει επέλθει μια σημαντική αλλαγή στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κυρίως λόγω της ε, διαχείρισης και της διακυβέρνησης από το, ε, του ΕΦΣΥ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Υπάρχουν πολλές νέες ε, δραστηριότητες έχουν διευρυνθεί οι εντολές διαχείρισης εκ μέρους της Κομισιόν και συμβουλευτικής υποστήριξης. Αυτή είναι μια τεράστια εξέλιξη στις δραστηριότητες τράπεζας που δεν πρέπει να παραβλέψουμε. Και τρίτον, όπως πάντα, υπάρχει αυτή η προσδοκία ότι η τράπεζα θα πρέπει να παρέχει προστιθέμενη αξία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακαιρεότητα, διαφάνεια και λογοδοσία. Πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα ε, όσον αφορά τα θέματα αυτά. Βάσει αυτών των τριών κριτηρίων λοιπόν, εγώ θα σας καλούσα ε, με την έκθεση αυτή να αναγνωρίσετε τα επιτεύγματα και τα προβλήματα. Όσον αφορά τα επιτεύγματα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η τράπεζα έχει ουσιαστικά επιτύχει τον οριζόντιο στόχο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. που αντιστοιχεί ο στόχος στο 30% επιτυγχάνοντας αξία 29,6% των στοχευμένων επενδύσεων. Κάτι για το οποίο εμεί κάνουμε έκκληση εδώ και καιρό. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν και να πνέσουμε την τραπεζά για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει σε αυτό το τομέα. Επιπλέον έχουμε τους κλιματικούς στόχους. Έχουμε τα κλιματικά ομόλογα, τα ομόλογα κλιματικής ευαισθητοποίησης, τα οποία έχουν εκδοθεί αυτό επηρεάζει τα περιβαλλοντικά θέματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό είναι μια άλλη εξέλιξη που πιστεύω αξίζει ε, να επενέσουμε. Τρίτον, έχουν γίνει προσπάθειες ε, ταχεία συμβολή ε, στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων μετανάστευσης και βιώσιμης ανάπτυξης με την έναρξη ομολόγων ε, ευαισθητοποίηση σε θέματα βιωσιμότητας. Και τρίτον, η Ελεγκτική Επιτροπή έχει συμπεράνει ότι τα οικονομικά της τράπεζας το ισοζύγιο της τράπεζας για το 2017 παρουσιάζει μια σαφή έκθεση για την οικονομική θέση της τράπεζας από την 31η Δεκεμβρίου του 2017 και τα αποτελέσματα των ταμιακών ροών και των δραστηριοτήτων της. Πέμπτον, υπάρχει η ενίσχυση της επίδοσης ε, εντός της ΕΤΕΠ ε, ένα συνεχές θέμα, πολύ σημαντικό. Διότι σαφώς η αλλαγή των δραστηριοτήτων της τράπεζας απαιτεί αντίστοιχες αλλαγές στο φιλοσοφία επίτευξη αποτελεσμάτων και πρέπει και εκεί να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Έκτον, θα πρέπει επίσης ε, να επισημανθεί δεν υπάρχουν ε, εγγύσεις όσον αφορά σε περίπτωση αποτυχίας ε, ε, κάποιων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΦΣΥ. Απαιτείται εδώ επαρκής, ε, έχει, γίνει, έχει υπάρξει επαρκής μέρημνα και διαχείριση κινδύνου. Επιπλέον υπήρξε βελτίωση της διαφάνειας μέσω της δημοσιοποίησης των αποφάσεων της Επιτροπής Επενδύσεων ΕΦΣΥ και, τα έγγρα, και των εγγράφων που έχουν εθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τα πρακτικά. Και αυτό είναι κάτι που είχε ζητηθεί εδώ και χρόνια και ε, αναμενόταν και για πάλι και πάλι πιστεύω ότι και εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες της τράπεζας. Τέλος 8 το 2017 η τράπεζα άρχισε να δημοσιοποιεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων και συγκρούσεων συμφερόντων και Διάφορε προφορές για τα έργα όπως εκτιμήσεις επιπτώσεων και περιβαλλοντικές εκτιμήσεις. Αυτά πιστεύω αξίζουν τον έπαινό μα. Δείχνουν ότι υπάρχει βούληση δράση, όχι μόνο βούληση, ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις προσδοκίες και ως απόκριση στις ε, μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά ζητήματα που μας απασχολούν και που αναφέρουμε σε αυτή την έκθεση 8 κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές και που παραμένει σημαντική ανισορροπία κατά την άποψή μου το γεγονός ότι τα μισά κράτη-μέλη έχουν λάβει το 80% των επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ τα άλλα μισά το 10%. Επίση υπαρχουν υπάρχουν τρία κράτη-μέλη τα οποία αντίστοιχα έχουν λάβει 16, 15 και 11% του συνολικού, της συνολικής αξίας. Το ίδιο συμπεραίνουμε όσον αφορά τη στρατηγική επένδυση στα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Και εδώ το Ευρωπαϊκό Συγγνώμη, Ταμείο ε, Στρατηγικών Επενδύσεων και εδώ έχουμε την ενδεικτική σύσταση, την ενδεικτική σύσταση γεωγραφικής συγκέντρωσης ότι 45% τριών μελών για να λάβουν τη συνολική επένδυση και αυτό που δεν πιστώσαμε είναι ότι αυτό που συνέβη είναι ότι τρία κράτη-μέλη ε, έλαβαν 47% ε, του συνολικού ποσού που υπογράφηκε το 2017. Κάτι δηλαδή στο οποίο εμείς εφιστούμε την προσοχή γιατί είναι δυσάρεστη η κατάσταση. Μετά Ήθελα επίσης να υπογραμμίσω κάτι. Έχουμε απευθύνει έκκληση για ολοκληρωμένη λεπτομέρη και εναρμονισμένη έκθεση των δραστηριοτήτων με αναλύσεις των επενδύσεων που έχουν εγκριθεί υπογεγραμμένων ε, των πόρων, των δικαιούχων, των τομέων και, των αποτελεσμα... και της ανάλυσης αποτελεσμάτων εξ όσον αφορά τις επενδύσεις. Έχουμε ένα τεράστιο εύρος διαφόρων εκθέσεων, ορισμένες ε, περισσότερο ότι έχουν κάποιες που έχουν εκδοθεί ενημερωτικά, κάποιες άλλες ως ε, στο πλαίσιο δημοσίων σχέσεων, αλλά δεν έχουμε συνολική ενιαία έκθεση που να τις συγκεντρώνει όλες μαζί με τρόπο σαφή, αναλυτικό και συγκεκριμένο. Αυτό, κατά την άποψή μου, παραμένει σημαντικό έλλειμμα των εργασιών ε, προβολή των δραστηριοτήτων τη Τράπεζα. Uh, Κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω είναι η συμπληρωματικότητα, η προσθετικότητα. Σε ποιο βαθμό δηλαδή η δράση της ΕΦΣΥ πραγματικά προσθέτει επενδύσεις σε ε, έργα που δεν θα ήταν ελκυστικά ή ε, σε άλλο πλαίσιο. Και εδώ πιστεύω ότι εξακολουθεί να υπάρχει αρκετά μεγάλο περιθώριο να εξετάσουμε προσεκτικά τα κριτήρια ε, καθορισμού ε, αυτού του παράγοντα και να δούμε κατά πόσο γίνονται οι δράσεις καθαρά εμπορικά ή κατά πόσο τηρείται αυτή η αρχή της προσθετικότητας. Επίσης ήθελα να αναφέρω οι διαδικασίες έγκρισης πιστώσεων και οι σχετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων χρειάζονται ολοκληρωμένη αναθεώρηση και ανανέωση ουσιαστικά. Όπως φαίνεται δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις σημερινές επιχειρησιακές ανάγκες σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της, του Ελεγκτικού Συμβουλίου της ε, Τράπεζας. Αυτό βρήκε η Ελεγκτική Επιτροπή της Τράπεζας και πιστεύω ότι αυτό χρήζει της προσοχής μας και περαιτέρω προσπαθειών επιπλέον σύμφωνα με την ίδια έκθεση φαίνεται να εξακολουθεί να είναι αδύνατη η αντιμετώπιση ε, η τήρηση κάποιων υπευθυνοτήτων και συνδυασμών που υπάρχουν ε, για διάφορες δραστηριότητες πρώτης και δεύτερης γραμμής. Εδώ θέλω να υπενθυμίσω τη σύσταση του Ombudsman του Δεμεσολαβήτη ότι είναι αναγκαίο να αλλάξει ο κώδικας διοντολογίας το συντομότερο δυνατόν ώστε οι αντιπρόεδροι να μην είναι επιφορτισμένοι με δράσεις στα ε, οικεία τους κρατημέλη. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, όπως κάνω πάντα, στο γεγονός ότι ακόμα αναμένουμε από την Τράπεζα συγκεκριμένες απαντήσεις όσον αφορά συστάσεις που έχουμε κάνει σε προηγούμενες εκθέσεις να επισημάνω τρεις τέτοιες, ε, τρία τέτοια αιτήματά μας σαφή υποβολή εκθέσεων για τα αποτελέσματα των επενδύσεων και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί δεύτερον πρόληψη των συγκρούσεων συμφορώντων που ανέφερα και διαφάνεια όσον αφορά τους ενδιάμεσους και τελικούς παραλήπτες των κονδυλίων, ειδικότερα όσον αφορά θέματα φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και διαφθοράς. Σας ε, έγραψα πιστεύω λοιπόν μια έκθεση η οποία σα δίνει μια πολύ σαφή εικόνα και ισορροπή εικόνα του τι γίνεται όσον αφορά τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του 2017 για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα έκθεση για τα θέματα που θέσατε. Είναι πολύ θετικά. Ο συνάδελφος Deutsch, παρακαλώ, από τους Σκιώδης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον κύριο Πυρίνσκι για τη δουλειά του που ήταν τόσο διεξοδική και σύνθετη. Και η προφορική του παρουσίαση. Λοιπόν, δύο πράγματα θα αναφέρω. Η, πρώτον, η ετήσια έκθεση και το κεφάλαιο 6 για το επενδυτικό ταμείο εξετάστηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο και κυρίως εις ό,τι αφορά την ε, ρύθμιση εντοπίστηκαν κάποιες ελλείψεις και αδυναμίες και αναφέρονται και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες πρέπει να γίνουν έλεγχοι από τις εθνικές αρχές ελέγχου. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν ε, είχαν την αρμοδιότητα και έτσι οι νομι... Ε, ε, ενώ θα έπρεπε να προβούν σε έλεγχο νομιμότητα των συναλλαγών εντοπίζω μία αντίφαση μεταξύ των δύο αυτών θεμάτων. Δηλαδή ε, θα έπρεπε ε, για να πάρουν χρήματα να είναι μήμιε. Κάποιες δεν ήταν. Σε πολλές περιπτώσεις οι δικαιούχοι επήραν κονδύλια που δεν θα έπρεπε γιατί είναι σε άλλο πεδίο δραστηριοτήτων. Στο 1 τρίτο των περιπτώσεων ε, κονδύλια δόθηκαν παράτυπα. Καλό θα ήταν η έκθεση αυτή με την τελευταία του εκδοχή να αναφέρει ότι πρέπει να δούμε αν το πολυνομοσχέδιο, το Omnibus, μπορεί να διασφαλίσει τις υποχρεώσεις που πρέπει να υπάρχουν και να εγγυάται και την σωστή εκτέλεση των προγραμμάτων ε, και τους σωστούς παραλήπτες. Και άλλη φορά είχαμε συζητήσει για αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να καταθέσω μια τροπολογία. Πρόκειται για το εξής. Μετά το Brexit, στο μέλλον θα έχουμε ένα θεσμικό όργανο με διαφορετική σύνθεση. Αυτό είναι σημαντικό αφενός και βέβαια αφετέρου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στην Βαλκανική. Πρόκειται για μια περιφέρεια πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό η δραστηριότητα της ΕΤΕΠ πρέπει να ενισχυθεί. Στις χώρες ΑΚΕ οι αιτίε της μετανάστευσης πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό είναι ένα, μια σημαντική συνιστόσα της δραστηριότητα της τράπεζας. Αλλά στα Δυτικά Βαλκάνια δεν είναι αρκετά μεγάλη η δραστηριότητα της τράπεζας, κυρίως σε σύγκριση με τις χώρες ΑΚΕΠ. Θα υποβάλω σχετική τροπολογία και καλό θα ήταν να ενσωματωθεί στην έκθεση. Μεγαλύτερη λοιπόν δραστηριοποίηση της ΕΤΕΠ στα Βαλκάνια. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Καντ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την αναγνώριση των όσων εμείς πετύχαμε, γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά στην ΕΤΕ. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια από τα θέματα που έχουν θίξει και να σας πω ότι και διμερώς θα μπορούσα να σας απαντήσω σε κάποια θέματα τα οποία θέλετε να δούμε. Για το θέμα το κατά πόσο μπορούμε όλα τα κράτη-μέλη να τα καλύψουμε, δηλαδή για το θέμα της γεωγραφικής κάλυψης, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως η ΕΤΕ δεν λειτουργεί με ποσοστό χωρών, αλλά βεβαίως προσέχουμε ιδιαίτερα να καλύψουμε όλα τα κράτη-μέλη. Και βεβαίως ε, πρέπει να το ετηθεί κανείς, αλλά θέλουμε να παραδώσουμε αυτό που επιθυμούν όλοι οι μετοχή μας. Να σας πω πως από όλους τους αριθμούς οι δικές μας ε, πράξεις και αυτές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων είναι σύμφωνα με τα όσα θέλαμε για το 2015, αλλά αν κοιτάξει κανείς ε, το ΑΕΠ ανακράτος ή το κατακεφαλήν, θα δείτε πως τα μικρότερα κράτη-μέλη όντως ευνοούνται από την ε, ε, ε, χρηματοδότηση της ΕΤΕ και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ κυρίως στην Ελλάδα, την Ιστονία, τη Βουλγαρία και τη Φιλανδία. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Έχουμε πάρει το θέμα αυτό πάρα πολύ σοβαρά και τον Νοέμβριο του 2018 επιβεβαιώνω πως υπάρχει αυτή η θετική τάση προς γεωγραφική διαφοροποίηση και στα πλαίσια του επενδυτικού ταμείου για το κομμάτι των τεχνολογικών επενδύσεων να σας πω πως σε, απόλυτα, σε απόλυτες τιμές Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία είναι το 46,8% κάτω δηλαδή από το όριο. Για τα Βαλκάνια να πω πως υπάρχει το θέμα της οικονομικής ανθεκτικότητας αυτό γιατί γνωρίζουμε πως πρέπει να κάνουμε παραπάνω πράγματα. Αυτή λοιπόν είναι η πρωτοβουλία μας που είναι συγκεκριμένη και όπως και άλλες ε, στιάζεται στα Δυτικά Βαλκάνια και με μεγάλη χαρά θα στείλουμε και περισσότερες πληροφορίες για το τι κάνουμε ε, και τι έχουμε στα σκαριά. Το σχόλιο που έγινε για το θέμα των αμυντικών επενδύσεων. Εμείς αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη πάρα πολύ σημαντικά και στα πλαίσια της χρηστής διαχείρισης και θα δούμε τι θα γίνει και με την έλλειψη κεφαλαίου λόγω Brexit. Θα δούμε την διαχείριση σε επίπεδο μετόχων για να δούμε ποιες είναι οι βελτιώσει που πρέπει να κάνουμε, συγγνώμη δεν ήταν αμυντικά κονδύλια, ήταν η γραμμή άμυνα. Να δούμε λοιπόν και για τη γραμμή άμυνα τι μπορούμε να πετύχουμε. Και βέβαια θα επιστρέψω για κάποια από τα άλλα θέματα τα οποία δεν μπορώ να απαντήσω σήμερα, αλλά σας υπόσχομαι πως θα το κάνω. Εμείς περιμέναμε να αποφανθείτε και επί της εκθέσεως πυρήνσκη θέματα ε, αντιφάσεων και συγκρούσεων και πότε... Θα υπολογίζουμε σε μια ακόμη ενημέρωση του Κοινοβουλίου. Um, we are partly, in a sense, already replying. Ε, ήδη απαντάμε. Υπάρχουν κάποια εκκρεμή θέματα τα οποία συζητούνται στο Συμβούλιο μας και όταν καταλήξουμε, ε, όπως στη γραμμή άμυνας, οπωσδήποτε θα επανέλθουμε στο Κοινοβούλιο. Αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε και τις εσωτερικές διαδικασίες της ΕΤΕΠ. Δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολείται και με τη σύγκρουση συμφερόντων των αντιπροέδρων όταν δραστηριοποιούνται στα κράτη-μέλη. Αυτό πότε θα ε, το συζητήσουμε. Επιβεβαιώνω ότι η σύγκρουση συμφερόντων συζητείται ως μέρος της μεταρρύθμισης της διακυβέρνησης και αφορά και για την ε, αντικατάσταση κεφαλαίων θα συζητηθεί και δεν θα καθυστερήσουν περισσότερο από το 2019. Καλώς. Θα θέλαμε ένα γραπτό σημείωμα σε σχέση με την γνώμη το, το, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε σχέση με την έκθεση Πυρίνσκη. Να σας πω το εξής. Γιατί ακούσαμε αυτές τις πολύ καλές ε, πληροφορίες που μας δώσετε στο καινούριο InvestEU. Θα ήθελα να μου πείτε τι άποψη έχει η τράπεζα αν με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η θέση της ως Ευρωπαϊκή Τράπεζα ή αν έχουν κάποιες επιφυλάξεις και θα ήθελαν ε, μεγαλύτερο αριθμό ε, τραπεζών στο Invest EU και όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν εσείς αυτό πώς το αντιμετωπίζετε. Η τράπεζα χαίρεται για τον ανταγωνισμό. Θα είστε εσείς οι πρώτοι που θα χαρείτε για τον ανταγωνισμό. Θέλετε να αντιδράσετε, να απαντήσετε σύντομα. το InvestEU πράγματι βρίσκεται υπό συζήτηση. Υπάρχουν διάφορες ε, αλλαγές σε σχέση με το ΕΦΣΥ. Όπως θα συμφωνήσουμε πιστεύω όλοι ε, έχουν στεφθεί με επιτυχία προς το παρόν. Συμφωνήσαμε με τα κράτη-μέλη για περαιτέρω συζητήσεις με την Κομισιόν ώστε να ληφθεί υπόψη και η δική μας ε, ε, εμπειρία ως τράπεζας, ώστε να είναι επιτυχή τα αποτελέσματα στο πλαίσιο του InvestEU όπως και έγινε και με το ΕΦΣΙ και συνεργαζόμαστε τώρα με την Κομισιόν για κάποια συμβιβαστική λύση που θα μας βοηθήσει να καθησυχάσουμε και κάποιους συνδυασμούς που υπάρχουν για την πρόταση InvestEU. Η Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ ζητεί το λόγο. Do wish to take the floor? Uh, I think it's me. να πάρει το λόγο, εγώ νομίζω. Ήθελα να επιβεβαιώσω αυτό που είπε η συναδελφός μου, ότι πράγματι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ ΕΤΕΠ και Κομισιόν για να βρεθεί μια συμβαστική λύση. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, αλλά σε αυτό το στάδιο η απάντησή σας δεν ε, βοήθησε. Εν πάση περιπτώσει θα επανέλθουμε. Ο εισηγητής θέλει το λόγο. Κύριε Πυρίνσκι, θέλετε να λάβετε πάλι το λόγο. Ναι, θα ήθελα. Ε, I thank, ε, my colleague, Mr. for... Να ευχαριστήσω λοιπόν και τον συνάδελφο κύριο Ντότς για μια από τις παρατηρήσεις του και για, την, για τον σεβασμό των υποχρεώσεων για τις μικρομεσαίες. Αλλά επίσης να σας πω πως ε, για τα Δυτικά Βαλκάνια συμφωνώ απόλυτα για τους προφανείς λόγους, για τους οποίους αναφερθήκατε και εσείς. Κυρία Πρόεδρε, έχω και εγώ τις ίδιες προσδοκίες με εσά πως οι εκπρόσωποι της τράπεζας θα είχαν την καλοσύνη να σχολιάσουν την έκθεση. Η απάντηση που έδωσε η κυρία, όπως την είπατε από την ΕΤΕΠ, είναι κάπως περίεργη. Γιατί το κεντρικό ζήτημα το οποίο εμείς και πάλι έχουμε θέσει είναι η γεωγραφική κατανομή. Και άκουσα αυτή την κλασική απάντηση ότι είναι το κατακεφαλήν, είναι το κατά που χρειάζεται. Δεν καταλαβαίνει η τράπεζα πως έχει κληθεί να φέρει τη συνοχή. Και υπάρχουν προφανέστατα περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε υποεπενδύσεις και που χρειάζονται τεράστιε επενδύσει για να ξεπεράσουμε τι ε, όλο και πιο βαθιέ ανισότητες και διαφορές οι οποίες απειλούν την ίδια την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ τώρα ακούω πολύ συντηρητικά και μπλαζέ σχόλια για το ότι αυτό επιθυμούν τα κράτη-μέλη, ότι εμείς προσπαθούμε να υπηρετήσουμε καθένα κράτος μέλος. Αυτό είναι τελείως απαράδεκτο, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον ως θέση της τράπεζας, γιατί είναι το κεντρικό ζήτημα που μας απασχολεί. Και μετά Μιλήσατε κι εσείς για κάτι το οποίο θα ήθελα και πάλι ε, να υπογραμμίσω που είναι η σύγκρουση συμφερόντων. Και εγώ δεν μπορώ να δεκτώ ως ε, εξήγηση κάτι το οποίο λέει πως στα πλαίσια ε, της ε, δεν συζητήθηκε το θέμα αυτό. Γιατί το θέμα αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στην πρώτη γραμμή, γιατί έχει να κάνει και πάλι με τη γεωγραφική κατανομή κονδυλίων. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αντί να καθυστερούμε, θα πρέπει η ΕΤΕ να παρουσιάσει στεναρή και ταχύτατη δράση. Δεν θέλω τώρα εγώ να ξανακνευρίζομαι. Θέλω να σας καλέσω. Αν έχετε την καλοσύνη να στείλετε γραπτά σχόλια για την έκθεση, το έχετε κάνει στο παρελθόν. Δεν θέλω να μείνω με την εντύπωση πως έχετε χάσει πια το ενδιαφέρον σας για το τι λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επειδή φτάνουμε στο τέλος της θητείας μας. Θα έχουμε καινούργια θητεία, θα έρθει άλλο κοινοβούλιο και θα είμαστε ακόμα πιο ισχυροί. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να το λάβετε υπόψη. Εντάξει, θα περιμένουμε τη γραφτή γραπτή γνωμοδότηση. Τελειώσαμε. Γιατί πρέπει να βιαστούμε, έχουμε άλλα τρία θέματα. Πρέπει να ε, ολοκληρώσουμε. Δεν έχω τίποτα άλλο εκτός από αυτά. Μια ε, φτάσαμε στο σημείο 7. ειδική έκθεση εκθέση -18 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Απαλλαγή 17. Ο κύριος ε, Νέβεν Μάτες από το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για αυτό το προληπτικό να του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ε, συγκεκριμένα αν το εκτελεί με τρόπο τέτοιο η Κομισιόν ώστε να επιτελέσει το σύμφωνο το βασικό του στόχο. Η Κομισιόν έχει πολλές αρμοδιότητες και διακριτική ευχέρεια κατά την εκτέλεση και κατά τη λήψη επιμέρους αποφάσεων όταν αποκτά τέτοια εξουσία. Το θεμητό ερώτημα είναι αν χρησιμοποιεί την εξουσία αυτή με τρόπο τέτοιο ώστε ο στόχος του κανονισμού να εξυπηρετείται. Θα έλεγα όχι. Και να εξηγήσω γιατί. Ποια ήταν η βασική ιδέα του προληπτικού βραχίων ήταν το εξής τα κράτη-μέλη έπρεπε να επιτύχουν το μεσοπρόθεσμο στόχο σε εύλογο διάστημα. Ο χρόνος δεν είχε εξειδικευτεί, αλλά αναφέρθηκε ότι θα έπρεπε η σύγκληση να είναι μισό, μισό της εκατό κάθε χρόνο. Και αναφέρθηκε ότι αυτή η σύγκληση θα έπρεπε να είναι ταχύτερη για υψηλά, πολύ υπερχρεωμένες χώρες. Και αν συγκρίνουμε τα διάφορα στοιχεία της εποπτείας ε, η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος που αφορά το ίδιο το έλλειμμα και η, υπερβολική, διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για το χρέος και το προληπτικό α, βραχίωνα. Αυτό είναι το πιο λογικό από όλα τα μέτρα. Αν λοιπόν μείνουμε στο προληπτικό βραχίωνα και δούμε και το μεσοπρόθεσμο στόχο, η Κομισιόν δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και τη δυναμική του χρέους, γιατί θα είχε εστιάσει στον προληπτικό βραχίωνα. Γι' αυτό είναι τόσο άλλο άλλος αυτό. Τώρα, ποια είναι τα βασικά στοιχεία του κανονισμού. Ε, είναι αυτή η ετήσια σύγκληση ε, με μισό δεκατό. Περισσότερες προσπάθειες θα πρέπει να γίνονται από τα κράτη-μέλη ε, για να μην φτάσουν στο ανώτατο όριο του χρέους. Κυκλικές συνθήκες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, προσαρμογή για μεγάλες μεταρρυθμίσεις και επενδυτικέ ανάγκες, αλλά και για ασυνήθιστα γεγονότα. Υπάρχει μια αμφιλεγόμενη ρύθμιση στον κανονισμό που λέει ότι μπορεί τα κράτη να παρεκκλίνουν ε, το λέει κάπως διαφορετικά, παρακλίνουν πάντως εννοεί, με 0,25% κάθε χρόνο. Το θέμα είναι πώς θα το αυτό. Αυτό θα το δούμε αργότερα. Πώς όμως ερμηνεύσε η Κομισιόν όλα, όλες αυτές τις οδηγίες του κανονισμού. Για δείτε εδώ το γράφημα. Η πρώτη γραμμή δείχνει πόσο γρήγορα η χώρα φτάνει από το έλλειμμα του 3% στο 0 ισοζύγιο, αν έχει ετήσιο ποσοστό μισό τα Εδώ το 3% είναι η χώρα η οποία ας πούμε βγήκε από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και βλέπετε με το μισό το 100 έχουμε σε 6 χρόνια 0 έλλειμμα ή σε 5 χρόνια αν έχουμε το, χρησιμοποιήσουμε το μισό το 100 έλλειμμα. Εδώ έχουμε συν, καιρούς όχι σε περίοδο κρίσης Συνήθι οικονομία. Με το μισό τα εκατό έχουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Η Κομισιόν όμω είπε ότι οι χώρε ε, παρεκκλίνουν μονίμως κατά μισό τα εκατό. Όχι μόνο δύο συνεχόμενα έτη και μετά δύο άλλα συνεχόμενα και μετά α, τρίτη φορά και μετά ε, άλλα δύο. Πάμε στα 12 χρόνια. Οπότε χρειάζεται έξι χρόνια είπαμε για το μηδενικό. Και τώρα ε, οι διάφορες εκπτώσεις. Υπάρχουν εκπτώσεις γιατί άμα γίνονται ε, μεταρρυθμίσεις και για τις επενδύσεις επίσης. Μπορεί να ε, έχουν έκπτωση 0,75% του ΑΕΠ. 3%, 3, χρόνια δηλαδή. Τώρα δεν είμαστε στα 12 χρόνια. Πάμε στα 15 χρόνια πια. Τώρα, αν γίνει κάποια, κάτι ασυνήθιστο, δεν υπάρχει εδώ ε, όριο, ξέρετε τι έχει εγκρίνει η Κομισιόν. Η Κομισιόν έχει εγκρίνει μισό της εκατό σε μια χώρα, σε σωρευτική βάση, οπότε έχουμε άλλα δύο χρόνια. Οπότε πάμε στα 17 χρόνια, έχουμε φτάσει ήδη στα 17. Στα 17 χρόνια όμως μπορεί να προκύψει και ύφεση βαθιά. Σε βαθιά ύφεση το διαρθρωτικό ισοζύγιο μέχρι τώρα πάντα επιδεινωνόταν. Δεν μιλάω για τη μεγάλη ύφεση μετά το 2008. Ας δούμε μια ήπια ύφεση το 2000. Εκεί επιδεινώθηκε το διαρθωτικό ισοζύγιο κατά 1,2% του ΑΕΠ. Οπότε προστίθενται εδώ άλλα πέντε χρόνια. Πάμε στα 22. Στα 22 χρόνια θα είμαστε ακόμα εδώ. Και επίσης η Κομισιόν ε, ε, ε, έχει ένα περιθώριο εκτίμησης και υπάρχει μια γενική ρήτρα που λέει η Κομισιόν ότι μπορεί να λάβει υπόψη τους λεγόμενους λοιπούς παράγοντες. Πώς θα λειτουργήσει αυτό σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Αυτό είναι μια ερώτηση και έχουμε και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιτευχθεί ο στόχος και αυτό αντιβαίνει σε αυτό που ορίζεται ως ο βασικός στόχος του κανονισμού. Είπα, εδώ είναι κανονική καιρή, όχι καιρή κρίσεων. Είπα ότι ο κανονισμός επίσης ζητάει περισσότερες προσπάθειες από υπερχρεωμένες χώρες. Λοιπόν, οι υπερχρεωμένε χώρε πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα και η Κομισιόν έχει μια μήτρα που τοποθετείται κανεί από το που είναι πούμε, στον επιχειρηματικό κύκλο. στι υποχρεωμένε χώρε πρέπει να γίνονται περισσότερα. Στι περισσότερε από αυτές τις κατηγορίες η Κομισιόν ζητάει 0,25% ε, παραπάνω. Εντάξει. Αλλά και έχουμε και φυσιολο... στους φυσιολογικούς ψάχνει, πάει, ζητάει μόνο 0,1%. Γιατί 0,1% στις ε, καλέ εποχέ και στι κακέ εποχές 0,25% και στι καλέ πάλι 0,25%. Αυτή η προϋπόθεση για τις υπερχρεωμένες χώρες στις κανονικές εποχές ε, είναι επαρκής. Έχουμε όμως ε, και αυτό το θέμα των εκπτώσεων όταν γίνονται επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Όταν η Κομισιόν μίλησε για την έκδοση για τις μεταρρυθμίσεις, αυτό ήταν καλό, γιατί δεν θέλαμε ε, δημοσιονομικοί περιορισμοί να επηρεάζουν την εφαρμογή, την εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων. Η μεταρρύθμιση έχει ένα κόστος συγκεκριμένο. Εμείς προτιμούμε να γίνουν όμως οι μεταρρυθμίσεις. Τότε όμως ε, περιορίζεται η ε, επιδείνωση το κόστος μόνο της ίδιας της μεταρρύθμισης. Η Κομισιόν, υποστηριζόμενη από το ΕΚΟΦΗΝ, είπε ότι δεν είναι το πραγματικό κόστος της μεταρρύθμισης που μετράει, αλλά η διάταξη πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός κινητροδότησης της μεταρρύθμισης. Οπότε όχι μόνο το παρόν έτος, το, το τρέχον έτος όπου γίνεται η μεταρρύθμιση, έχουμε το κόστος και μειώνουμε την ανάγκη για προσαρμογή, αλλά οι δαπάνες επεκτείνονται και στα επόμενα χρόνια. Αυτό αντιβαίνει στο πνεύμα του κανονισμού, θεωρούμε εμείς. Επίσης, το ίδιο ισχύει για την έκπτωση για τις επενδύσεις. Γιατί δεν, ζητάμε, δεν ζητάει εδώ να αυξηθούν οι επενδύσεις σε ένα συγκεκριμένο έτος σε σχέση με το ΑΕΠ. Όχι, λέει, ε, είναι αρκετό να, να, να αυξηθεί ονομαστικά γιατί σε σχέση με το ΑΕΠ μπορεί να μειωθεί κιόλα. Ένα έτος. Τα επόμενα έτη όμως, ό,τι πάρουμε για αυτό το έτος, μεταφέρεται. Δηλαδή η έκπτωση μπορεί να γίνει για οτιδήποτε. Μπορεί να σταματήσουν οι επενδύσει, αλλά να ωφελείστε από την έκπτωση για λόγους επενδύσεων, για να γίνονται επενδύσεις. Και το ίδιο ισχύει για τα απρόβλεπτα, τα εξαιρετικά γεγονότα. Γιατί όχι μόνο ε, περιοριζόμαστε στο χρόνο που θα γίνει, αλλά δημιουργείται μια βάση, θεμελιώνουμε αν θέλετε, να δικαίωμα και για τα επόμενα χρόνια. Έτσι ε, έχει το θέμα και δεν, δεν σχολιάζω άλλο. Επίσης, άλλο σημαντικό, η Κομισιόν χρησιμοποιηθεί την συμμόρφωση με τον προληπτικό βραχίον ως επιχείρημα για να μην αρχίσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, γιατί δεν μειώνει το χρέος η χώρα. Όμως η Κομισιόν λέει ότι το διαρθρωτικό ισοζύγιο επιδεινώνεται σε υπερθερωμένες χώρες. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρεί ότι αυτό είναι αρκετό στο βαθμό που ευθυγραμμίζεται με όλα τις εκτόσεις ότι αυτό είναι αρκετός λόγος για να μην αρχίσει η διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος με βάση αυτό το κριτήριο. Και τι γίνεται στην πραγματικότητα. Βλέπετε λοιπόν ότι το ε, διορθωτικό ισοζύγιο μετά το 2014 σταμάτησε να βελτιώνεται. Μετά υπήρχαν πιέσεις ε, από τις αγορές, ε, βελτιώνονται, κάνουν προσπάθειες οι χώρες, βελτιώνεται το διορθωτικό ισοζύγιο, μετά σταματάει. Ο μέσος όρος δεν μετράει. Σε μέσο όρο, εκφρασμένο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει καλά. Αλλά ε, η αλυσίδα δεν ε, κρίνεται από τον πιο δυνατό κρίκο, αλλά από τον πιο ασθενή. Τι γίνεται λοιπόν με τις υποχρεωμένες χώρες εν προκειμένου. Εδώ βλέπετε τι απαιτήθηκε να κάνουν οι υπερχρεωμένες χώρες μετά το 2013 όταν άρχισε η ανάκαμψη και ήταν αρκετά έντονη. Η μπλε γραμμή σας δείχνει τι ε, προέβλεπε η μήτρα αυτή της Κομισιόν και η κόκκινη γραμμή τι έκαναν τα κράτη. Η Ιρλανδία έκανε περισσότερα από τα απαιτούμενα. Όλες οι άλλες οι υπερχρεωμένες χώρες έκαναν λιγότερα. Και αυτό που εκπλήσει, ε, όχι εκπλήσει αλλά είναι ανομαλία, είναι ότι ε, το διαρθρωτικό ισοζύγιο 2014-2017 στην Ιταλία και Ισπανία επιδεινώνονται, δεν βελτιώθηκαν, επιδεινώθηκαν. Οπότε αυτές είναι υπερχρεωμένες χώρες. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Δεν έχει σημασία για άλλες χώρες τι κάνουν. Τι κάνουν οι άλλες χώρες δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία έχει τι κάνουν οι υπερχρεωμένες χώρες και τι γίνεται σε αυτές. Και βλέπετε εδώ το δίκτυ χρέου στι υποχρεωμένε χώρε. Βλέπετε ότι δεν υπάρχουν αλλαγέ εκτό από την Ιρλανδία. Σε όλε τι άλλε χώρε το ύψο του χρέου και ο δίκτυς χρέους ΑΕΠ παρέμεινε ο ίδιος. Αλλά αυτέ είναι χώρε που έχουν πάνω από 90% δείκτη χρέου, ΑΕΠ. Πολύ χρεωμένε. Είναι ενδιαφέρον να τις συγκρίνουμε με μέτρια χρεωμένες που έχουν ας πούμε, μεταξύ 60 και 90 δίκτυ χρέους. Εδώ, αυτές οι χώρες λοιπόν συμπεριφέρονται με ένα λογικοφανή τρόπο, με την έννοια ότι μετά την κρίση, αφού πέρασε η κρίση, οι δημοσιονομικές τους πολιτικές πάνε για να μειώσουν, ε, απευθύνονται στο να μειώσουν τον δίκτυο. Γίνεται αυτό. Στις πολύ υπερχρεωμένες χώρες δεν γίνεται όμως αυτό και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Και πάω στις συστάσεις. Είπαμε λοιπόν πρώτα απ' όλα πως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την απόκληση να τη λάβει υπόψη. Γιατί θα μπορεί το κράτος βέβαια να αποκλίνει ε, με κάποια ε, ελάχιστα ποσοστά ε, από τις απαιτήσει της. Αλλά μας είπε το board της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αυτό χρήζει αναθεώρησης. Και μετά έχουμε να δούμε και στο Matrix τι έχει πει ταυτόχρονα για το ποιοι θα είναι οι κανόνες για την περίπτωση της απόκλησης. Αν αυτή η απόκληση δεν είναι μόνιμη, τότε ίσως τα όσα έχουμε στο Matrix είναι αρκετά. Αν όμως δεχτεί πως αυτή η απόκληση μπορεί να συνεχίζεται αιωνίως, τότε θα πρέπει να αλλάξουν και τα νούμερα στο Matrix. Και αυτό θα είναι η δική μας σύσταση. Επίσης, για τις πολύ χρεωμένες χώρες, στους κανονικούς καιρούς θα πρέπει να υπάρχει ε, μια πιο ισχυρή υποχρέωση από την προσαρμογή που έχουμε αυτή τη στιγμή που είναι το 0,1%. Και είπαμε επίσης, ε, τα διορθωτικά μέτρα για το υπερβολικό έλλειμμα θα πρέπει να έχουν ε, δημιουργεί με έναν τρόπο που θα επιτρέπουν πως το... η διόρθωση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη δημοσιονομική ισορροπία, τη διορθωτική ισορροπία, έτσι ώστε να μην έχουμε υποδιόρθωση. Γιατί διαφορετικά, ε, πώς μπορεί το διορθωτικό σκέλος να είναι ε, λιγότερο στεναρό από το προληπτικό. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το σκέλος το διορθωτικό να μην είναι αδύναμο, ε, γιατί δεν μπορούν όλα να γίνουν σε επίπεδο προληπτικού σκέλους δεν δέχτηκε την πρώτη λύση που προτείναμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπε πως δεν χρειάζεται να σφίξουμε το τρέχον πλαίσιο. Αλλά κάποιες μικροσυστάσεις τις δέχτηκαν και τουλάχιστον αυτό μας ικανοποιεί. Πάντως θεωρούμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το δει διαφορετικά. Γιατί σε αυτό το συνδυασμό με το Matrix και τη δυνατότητα της μόνιμης απόκλησης πρέπει να σας πω ότι δεν γίνεται να έχετε το 0,5% σημείο αναφοράς και μετά να πείτε ναι, ένα κράτος όμως θα μπορεί από εδώ και στο εξή να αποκλίνει κατά 0,5%. Αυτό θα πρέπει να το ξαναδείτε. Επίσης, η ρήτρα αναθεώρηση θα πρέπει να συνδέεται απερίφραστα στο, με το κόστος μεταρρυθμίσεων και η ρήτρα για τις επενδύσεις, εάν θέλετε να τη διατηρήσετε, θα πρέπει να οδηγεί σε αύξηση ε, των επενδύσεων σε σχέση με το ΕΠ. Διαφορετικά πώς θα λειτουργήσει. Και βέβαια για, ε, για κάποιες έκτακτες, ε, έκτακτες πληρωμές θα πρέπει αυτό ζωρίτε να επιτρέπεται για ένα έτος και όχι να επεκτείνεται και στα επόμενα. Αυτές είναι οι συστάσεις μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Αν έχετε και άλλες ερωτήσεις, με χαρά να απαντήσω. Ja, vielen Dank, Herr Wir sehen, dass hier der ehemalige Notenbanker ganz offensichtlich in seinem Element ist. Φαντάζομαι ότι ε, είναι, ε, ε, είμαστε στο στοιχείο μας σε σχέση με τα, ε, προβλήματα που έχουν και οι τράπεζες. Ναι, ο κύριος Ναι, έχετε δίκιο. Συνήθως δεν είναι τόσο αναλυτικές οι παρουσιάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και αυτό πιστεύω είναι κατανοητό. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια ασυνήθιστη έκθεση για το ελεγκτικό συνέδριο αφορά ένα κέριο ζήτημα το πώς το, λειτουργεί το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα λειτουργεί υπερβολικά χαλαρά, λειτουργεί σωστά, λειτουργεί υπερβολικά συντηρητικά, διότι και αυτή την πτυχή δεν πρέπει να ξεχνάμε έχω μια μεγάλη παρουσίαση και μια μικρή τη έκθεση. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομο, διότι ο συνάδελφο Δε Jong έχει και άλλα δύο σημεία μετά. Θα προσπαθήσω ωστόσο να συνοψίσω τα όσα έχω καταλάβει εγώ από αυτή την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Η θεμελιώδης ε, λογική στην οποία βασίζεται το προληπτικό σκέλος είναι ότι με την επίτευξη ενός μεσοπρόθεσμου στόχου διαρθρωτικής ισορροπίας έχουμε τον καλύτερο τρόπο βιώσιμης ανάπτυξης των οικονομιών, επίτευξης ε, μεγαλύτερης απασχόλησης, ανταγωνιστικότητας κτλ. Αυτό πιστεύω είναι το βασικότερο ζήτημα στο οποίο βασίζονται ε, τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται στην έκθεση και οι απαντήσει τη Κομισιόν. Θέλω να επαναλάβω κάτι πολύ συνήθιστο ε, που παρατήρησα σε αυτή την περίπτωση. Όπως νομίζω ότι υπάρχει απόλυτη διαφωνία μεταξύ ελεκτικού συνεδρίου και Κομισιόν όσον αφορά το εξή ερώτημα. Λειτουργεί το προληπτικό σκέλος. Το συνέδριο το έχει πει σαφώ. Ω αποτέλεσμα της απομάκρυνσης ε, από το καταστατικό του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης κατά την εφαρμογή του σκέλους ε, δεν διασφαλίζει η Κομισιόν την επίτευξη του βασικού στόχου της σύγκληση των μεσοπρόθεμων στόχων σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η Κομισιόν επίσης είναι σαφής. Απαντά βάσει αντεπιχειρημάτων, εκτενών μάλιστα, ότι απορρίπτει το συμπέρασμα του Ελεκτικού Συνεδρίου ότι η Κομισιόν δεν έχει διασφαλίσει την επιτευξή του κύριου στόχου του κανονισμού. Πώς αποφασίζουμε ποιο έχει δίκιο και ποιο δεν έχει. Εγώ προσπάθησα να συνοψίσω όσο το δυνατόν πιο επιγραμματικά τα επιχειρήματα του Ελεκτικού συνεδρίου και πιστεύω ότι ουσιαστικά μιλάμε εδώ για πέντε βασικές διαπιστώσεις. Πρώτον, ο κανονισμός είχε κατάλληλη βάση για τη σύγκληση των μεσοπρόθεσμων στόχων, αλλά περιλαμβάνει διφορούμενες διατάξεις που επιτρέπουν μεγάλο περιθώριο απόκλησης. Υπάρχει λοιπόν κάποιο πρόβλημα με τον κανονισμό. Δεύτερον, η Κομισιόν έχει ασκήσει υπερβολικά τη διακριτική ευχαίρεια που της χορηγήθηκε, χωρίς ωστόσο να εστιαστεί στον κύριο στόχο τη μεσοπροθέσμης ισορροπίας, ε, μεσοσύγκλησης. Ε, υπάρχουν 5-6 επιχειρήματα που παρουσίασε ο κ. Μάτης για αυτό το θέμα στις διαφάνειες που μας έδειξε. Η μήτρα που ανέφερε, το, η απέτηση αυτή, δεν λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι η Κομισιόν δεν ε, ανέλησε κατά πόσο οι παράμετροι που περιέχει προσανατολίζονταν επαρκώ προ τον MTO, οι ρήτρε υλοποίηση και ευελιξία, έτσι όπω τι χρησιμοποιεί η Κομισιόν υπάρχουν καθυστερήσει ε, ε, το σωρευτικό αποτέλεσμα των ρητρών ευελιξίας και το περιθώριο απόκληση, εμποδίζει την επίτευξη του μεσοπροθεσμού στόχου περαιτέρω. Στο 4, η Κομισιόν έχει εισάγει ένα περιθώριο εκτίμησης που αναφέρεται και περιθώριο διακριτικής ευχέρειας που επίσης χαλαρώνει ε, την πειθαρχία στον όλο τομέα περαιτέρω και η τελευταία παρατήρηση του συνεδρίου είναι ότι δεν είχε δοθεί άδεια για υπερβολική ευελιξία Άλλες προσεγγίσεις υιοθετήθηκαν πολύ αδύναμες, πολύ, πολύ Αυτή είναι η επιχειρηματολογία για τη δεύτερη ε, δήλωση ότι ήταν υπερβολικά δύναμη εφαρμογή των κανόνων. Μετά, όταν πέρασε η κρίση, ήταν πιο χαλαρή η πίεση για την, εφαρμογή, για την επιδεύξη του στόχου και εκεί αποδυναμώθηκε η κατάσταση. Τέταρτον, υπάρχουν διάφορε τεχνικέ πτυχέ τη αξιολόγηση τη Κομισιόν που απαιτούν βελτίωση. Και τέλο, οι συστάσει τη Κομισιόν κυρίω ε, αφορούν καταστάσει ε, ε, ενίσχυσης της ανάκαμψης με αποτέλεσμα όμως ασύμετρα συμπεράσματα. γιατί χρειάζεται κάποια μέτρα να υπάρξουν τα οποία θα περιορίσουν τέτοιε αυξήσεις για λόγους ε, δημοσιονομικού ισοζυγίου. Ανέφερε κ. Μαθή λοιπόν τις διάφορες ε, συστάσεις που κάνει το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν θα απαριθμίσω τι απαντήσει της Κομισιόν, γιατί έχουμε εδώ εκπροσώπους της Κομισιόν, τον Διευθυντή, τον κ. Πέντς, ε, από το Τμήμα Δημοσιονομική πολιτική και μείγματο Πολιτικής, ο οποίο είμαι βέβαιο ότι θα θέλει να μα παρουσιάσει τι θέσει της Κομισιόν όλα αυτά, για όλα αυτά ε, στις διαπιστώσει του ελεγκτικού συνεδρίου. Και τέλος, οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου να είναι έξι, δεν θέλω να τις επαναλάβω, απλά θέλω να παρατηρήσω ότι οι βασικές ε, είναι οι εξής, ότι η Κομισιόν δεν τις δέχεται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το Matrix, με τη μήτρα. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ευελιξία. Η υλοποίηση του κανονισμού δέχεται ότι υπάρχει περιθώριο για καλύτερη πληροφόρηση και υλοποίηση. Και για προσαρμογή του διατακτικού. Θέλω να αναφέρω κάτι που αναφέρθηκε στην αρχή. σαφώ το ελεγκτικό συνέδριο επικρίνει την Κομισιόν για την υπερβολική τη ευελιξία. Εγώ από πλευρά μου αμφιβάλλω κατά πόσο είναι επαρκώ ευέλικτη η Κομισιόν. Διότι όπω αποδείχθηκε το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη έχει εξελιχθεί στο πιο περίπλοκο παγκοσμίω σύνολο κανόνων για διαχείριση κάποιου προπολογισμού και δεν είμαι βέβαιος ότι όλοι γνωρίζουν εδώ απολύτως σαφώς τι λένε. Παρατηρούμε εξελίξεις καθημερινά με τεράστιες διαφορές όσον αφορά την κατανόησή μας ε, αυτής της δεσμής μέτρων. Η επικρίση λοιπόν του ελεγκτικού συνεδρίου θεωρώ είναι μια καλή ευκαιρία να επανασχεδιάσουμε εκ βάθρων το... τη δεσμή μέτρων αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα, δύο λεπτά παρακαλώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που μου δίνετε το λόγο και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μάτες για την παρουσίαση που έκανε και συμφωνώ με όσα τα λένε. Αυτό που θα ήθελα, γιατί ίσως δεν το ξέρω, είναι να ρωτήσω το εξή. Είναι σαφές πως έχουμε ένα μάτριξ, ναι, θαύμα και θα λύσει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και για το έλλειμμα, και για το πλεόνασμα, γιατί όπως είπε και ο κύριος Μάτες υπάρχουν και κράτη όπου το υπερπλεόνασμα είναι πραγματικά πολύ κακό για όλους τους υπόλοιπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε μου, στο Matrix φαίνεται από πού προέρχεται το χρέος μιας χώρας γιατί, για την Ισπανία. Ξέρω και άλλους, αλλά για αυτούς που ξέρω, καταρχήν ήταν ιδιωτικό χρέος, το οποίο ξύνεται με τοξικά προϊόντα και παραπάνω από τοξικά από τις τράπεζες, γιατί αυτή τη στιγμή το λένε όλα τα δικαστήρια, και κάνουμε διάσωση τραπεζών με δημόσια χρήματα. Άρα λοιπόν αυτά τα ιδιωτικά τοξικά δάνεια έχουν γίνει δημόσια, κρατικά. Θέλουμε λοιπόν ένα είδος μάτρεξ για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που δημιούργησαν οι τράπεζες και τα ιδιωτικά δάνεια και χρέη. Αυτό το έχετε λάβει υπόψη. Και πείτε μου, το ελεγκτικό συνέδριο ποια έτη μελέτησε για να μας δώσει αυτό το μάτριξ και για να την ερμηνεύσει έτσι. Και μπορούμε να το εφαρμόσουμε όσο δεν έχουμε κρίση. Αλλά καταλαβαίνετε πως η κρίση του 8 ήταν η κρίση με κεφαλαία. Οπότε, ποια έτη μελετήσατε κύριε Μάτες για να μας δώσετε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό ήθελα να μάθω. Ο κύριος Σπέγκ από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να μην υπερβούμε το χρόνο. Αλλά είμαι διατεθειμένος να απαντήσω πιο λεπτομερείς ερωτήσεις αν χρειαστεί. Καταρχήν, Δύο πράγματα θα τονίσω στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και την παρέμβαση του κυρίου Μάτες του ίδιου. Στην αρχή της παρέμβασης του κύριος Μάτες ε, εστίασε στο αν η Κομισιόν χρησιμοποίησε τη διακριτική της ευχέρεια για να επιτύχει το στόχο του συμφώνου. Μόνο κάποια στιγμή αργότερα αναγνωρίζει ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα τα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου δείχνουν μια πλήρη σχεδόν συμφωνία μεταξύ Κομισιών και Συμβουλίου. Γιατί, όπως γνωρίζουμε, εν πολλής η, η εφαρμογή και η υλοποίηση του συμφώνου είναι επιμερισμένη αρμοδιότητα Κομισιών και Συμβουλίου. Ο καθένας στον τομέα του. Είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Ε, όταν μιλάμε για το, αυτό το Matrix, όταν μιλάμε τη μήτρα αυτή ή τη ρήτρα ευελιξίας, αυτά δεν είναι ιδέες που τις κατέβασε μονομερός η Κομισιόν και τα, τις πρότεινε τις επέβαλε στα κράτη-μέλη. Πρόκειται για διατάξεις που είναι λεπτομερέστατες και έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ σε κοινή θέση. Λοιπόν, αυτό μην το ξεχνάμε και υπάρχουν και λεπτομέρειες. Ε, δεν θα προλάβουμε να τα πω όλα. Τώρα το άλλο που επίσης υπογραμμίστηκε στην παρέμβαση του κυρίου Πυρίνσκι είναι ότι η παρατήρηση του ελεγκτικού συνεδρίου φαίνεται να απευθύνεται κάποιες φορές στην Κομισιόν, δηλαδή για το πώς ε, ε, υλοποίησε το σύμφωνο και είπα ότι πάνε μαζί η Κομισιόν Συμβούλιο, άλλες φορές φαίνεται να απευθύνεται η κριτική στον ίδιο τον κανονισμό. Αυτό που είπε ε, ομολογουμένος, αμφιλεγόμενη διάταξη στον κανονισμό. Έτσι είπε ο κ. Σπυρίνσκι. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε για πολλή ώρα σχετικά με το με την επόμενη διατύπωση ή την επόμενη τροποποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας. Αλλά τώρα το καθήκον μου στη Γενική Διεύθυνση και το καθήκον της Κομισιόν γενικότερα είναι να είναι πιστοί στο νόμο. Παράδειγμα, έχουμε αυτό το θέμα, το περιθώριο απόκληση που είναι χαμηλό και μια χώρα ε, θα πρέπει να προσαρμόζεται με κάποιο ρυθμό 0,5% ε, σημείο αναφορά. και μετά υπάρχει και ένα άλλο 0,25% περιθώριο απόκληση σε αιτήσια βάση και ε, αυτό αναφέρεται σε ειδική διάταξη του νόμου, του, του, συμφώνου δηλαδή. Και οι νομοθέτες, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, την εποχή εκείνη, είπαν ότι πρέπει να υπάρχει. Και αν ξέρετε από το τι πιστεύω προσωπικά για αυτή τη διάταξη, δεν είναι δουλειά της Κομισιόν ούτε να αγνοήσει, ούτε να καταστρατηγήσει αυτή τη διάταξη τεχνητά ε, αυξάνοντας το περιθώριο τα, τα, της ε, μάτρεξ, της μήτρας αυτής. Κατά τον ίδιο τρόπο το σύμφωνο ε, δεν ε, είναι αμετάκλητο. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση 2005 του συμφώνου. Δεν προβλέπει ότι οι εκπτώσεις για διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να περιορίζονται στο ε, δημοσιονομικό κόστος της μεταρρύθμισης αυτή. Μπορεί να είναι μια ερμηνεία, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ε, στο, στο νομοθέτημα. Ίσως αργότερα διατυπωθεί έτσι το σύμφωνο. Ε, υπάρχουν πολλές διαφορετικές ιδέες σχετικά με το στόχο του συμφώνου και ήταν πολύ χρήσιμο ότι ο κύριος Μάτες αφενός και ο κύριος Πυρίνσκι από την άλλη σας έδωσαν τις, τα δύο άκρα. Γιατί ο ένας είπε ότι η Κομισιόν ήταν υπερβολικά ε, ευέλικτη ή άκαμπτη και ο κύριος Σπυρίνσκι είπε η Κομισιόν ίσως δεν υπήρξε αρκετά ευέλικτη σε σχέση με το σύμφωνο. Θα έμπαινα στον πειρασμό να πω ότι είναι Μέντιο Στατ και εγώ είμαι στο κέντρο κρατώντας ίσες αποστάσεις και από τους δύο μπαίνω σε αυτό τον πειρασμό. Είμαστε πεπισμένοι ότι η εφαρμογή της ευελιξίας, ιδιαίτερα μετά από μία κρίση που ήταν εξαιρετικής φύσεως, πιστεύουμε ότι ήταν λογική και αναλογική λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση υπάρχουν επιμέρους ε, θέματα. Υπάρχει και η έκθεση της Ευρωπαϊκής ε, Δημοσιονομικής Επιτροπής που αναδεικνύει κάποια θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Πάντως, ε, περιορίζομαι στο στάδιο αυτό σε αυτές τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις και αν χρειαστεί ευχαρίστως να δώσω κάποιες επεξηγήσεις. Ο κύριος Μάτης. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως κατόπιν έλαβε την έγκριση του ΕΚΟΦΗΝ και για το Μάτριξ και για αυτές τις ευελιξίες. Όμως αυτό δεν είχε προβλεφθεί από τον κανονισμό. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να τα αποφασίζει, έλαβε αυτή την απόφαση, ξεκίνησε να εφαρμόζει το Μάτριξ και μόνο αργότερα έλαβε τη συγκατάθεση του ΕΚΟΦΗΝ. Τώρα, δικό σας θέμα να αποφασίσετε. Αν αυτό είναι εντάξει. Δεν υπάρχει κάτι στη διατύπωση του κανονισμού όπου για να εφαρμοστούν αυτές οι ευελιξίες και για την έγκριση των εφαρμοστικών κανόνων θα πρέπει να επιστρέψει στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι, οι υποχρεώσεις είναι οι γνωστές και τις κάλυψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν νομίζω ότι αυτό ήταν ιδιαίτερο χρήσιμο βέβαια με τα, μεταποτελέσματα που είχε, αλλά αλλά πρέπει να σου πω ότι οι περισσότερες χώρες συμπεριφέρονται καλύτερα από αυτό το οποίο απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι οι πολύ χρεωμένες χώρες οι οποίες ευνοούνται πιο πολύ από αυτή την εφαρμογή και την ερμηνεία των κανόνων που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τη μόνιμη δυνατότητα απόκληση. Ξέρετε πως το Fiscal Board της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε πως αν γίνεται αυτή η απόκληση θα πρέπει την επόμενη χρονιά να διορθώνεται. Και αυτό ήταν μέσα στις δυνατότητες τις ερμηνευτικές που είχε. Και δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και είχε τότε την δυνατότητα να ζητήσει και διευκρινήσει και προσαρμογή στον κανονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν λύνονται και το τι αποτείται και αν είναι αυτό το ε, ένα τέταρτο, το 0,25 με συγχωρείτε ή όχι. Η Matrix δεν χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια του διορθωτικού σκέλους, αυτό το Matrix. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο διορθωτικό σκέλος, και την εποχή της κρίσης. Η μεγάλη πλειοψηφία το έκαναν, οπότε το Μάτριξ εκεί δεν ήταν νομικά εφαρμοσιμό σε χώρες οι οποίες βρίσκονται σε προληπτικό σκέλος. Αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όχι μόνο χώρες που, στις οποίες αναφέρθηκα αλλά και κάποιες άλλες θεωρούσαν πως μπορούν να ξεφύγουν από το διορθωτικό σκέλος λόγω απλώς ε, κυκλικής βελτίωσης, παρόλο που δεν συμπίπτουν με τους μακροπρόθεσμους στόχους, δεν είναι οι χώρες που ανέφερε, ήταν κάποια άλλη. Οπότε λοιπόν, όπως σας είπα και εγώ, θα πρέπει αυτό το πλαίσιο να το ξαναδούμε και ίσως θα πρέπει να είναι κομμάτι του θεματολογίου στο μέλλον. Ευχαριστώ. Και θα συνεχιστεί η ιστορία αυτή με την Ιταλία, θα δούμε πρακτικά παραδείγματα και θα δείξει η ιστορία ποιος είχε δίκιο. Ελπίζω, ελπίζω να μην πάθουμε καμιά ζημιά όταν θα κρίνει η ιστορία ποιος είχε, ποιος είχε δίκιο και ποιος όχι. Ο κύριος Σπυρίνσκι. Κυρία Πρόεδρε, τέτοια ώρα και με τέτοια θερμοκρασία εδώ στην αίθουσα δεν νομίζω ότι θέλω να παρατείνω άλλο τη συζήτηση αυτή. Ε, προέκυψε από τη συζήτηση ότι τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι κέρια. Το μόνο που έχω να πω κλείνοντας ε, ήταν κάποια ερώτηση ουσιαστικά. Ο ενδιάμεσος ε, στόχος και ε, το Matrix φαίνεται να είναι σαν ιερία γελάδα. Δεν μπορεί να τα αγγίξει κανείς. Θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πάντα, αλλά πρέπει ανα πάσα στιγμή να τηρούμε αυτά καθημερινά αυτό εμένα με αφήνει γεμάτο απορίες γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία της ε, λιτότητας η οποία κατέρευσε, έχει αποτύχει. Ευχαριστώ. Ε, θα πάτε κύριε Μάτες να κάνετε αυτή την έκθεση στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Όχι ακόμα. Δεν έχετε κλείσει να πάτε. Θα έπρεπε να το κάνετε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Θα συνεχιστεί η αντιπαράθεση όμως. Πάμε στο σημείο 8 εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινή δήλωση που διασφαλίζουν το κοινοβουλευτικό έλεγχο των αποκεντρωμένων οργανισμών. Ο συντάξης γνωμοδότης είναι ο συνάδελφος Ντένις Δε Γιόγκ. Του ζητώ συγγνώμη που είχε να περιμένει τόση ώρα. Λοιπόν, να παρουσιάσει τη γνωμοδότηση ο κύριος Δε Γιόγκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μην ανησυχείτε, δεν με πειράζει που περίμενα. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τι συζητήσει που έγιναν, ε, ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσε. Θα είμαι σύντομο. Μιλάμε εδώ για μια μη νομοθετική γνωμοδότηση της Επιτροπής ΑΦΚΟ. Αυτή είναι η Επιτροπή τη ουσία. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο ουσιαστικά εδώ. Εδώ, σε αυτή την ε, Επιτροπή, έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό πάνω από μία φορές. Έχουμε συζητήσει το θέμα του IIWG και πάντα καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα ότι κάθε φορά που συζητάμε για το κατά πόσο η κατανομή των οργανισμών έχει γίνει με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο και όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους και τα και τα καθηκοντά τους πάντα ζητάμε από την Κομισιόν να μας δώσει αποδείξεις Κάθε κράτος μέλος έχει ένα διοργανισμού. Το κοινοβούλιο το έχει εξετάσει και στην IAWG δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε ιδιαίτερα λόγω έλλειψης προτάσεων σχετικών από την Κομισιόν. Εκεί υπάρχει κάποιο είδου διένεξη, διότι από τη μία πλευρά υπάρχει επιθυμία να επιληθεί το ζήτημα των τελών που ζητούν οι οργανισμοί. Εμεί θα προτιμούσαμε τα τέλη να πηγαίνουν στην Κομισιόν ώστε να παραμένουμε εμεί ε, ανεξάρτητοι. Να παραμένουν ανεξάρτητοι αυτοί που λαμβάνουν άδεια. Θα υπήρχε έτσι και μια οικονομική εισρωή ανεξάρτητη από τα τέλη. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο που είχα να αναφέρω εδώ στην γνωμοδότηση. Και μετά υπήρξε και μια ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Προέδρου του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν όταν ένας οργανισμός ε, μετακομίζει από μια χώρα σε μια άλλη το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει. Εμείς δεν συμμετείχαμε στη διαδικασία που οδήγησε στην επιλογή της νέας έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και αυτό το καλύπτω σε αυτή τη γνωμοδότηση. Τα υπόλοιπα είναι τα κλασικά πράγματα που πάντα ζητάμε ε, πιο απλοποιημένες, ε, ομογενοποιημένες εκθέσεις, συστάσεις. που έχουν γίνει από την διοργανική ομάδα εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς ε, να, να υλοποιούνται οι συστάσεις αυτές. Δεν είναι μεγάλη γνωμοδότηση. Είναι ιδιαίτερα σύντομη. Έχουμε συνεργαστεί στενά με τους σκιώδεις για όλα αυτά. Κυρία Κάντεμπαχ, παρακαλώ. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, τον κύριο Ντένις Διγιόγκ, Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Εδώ και χρόνια είχα να κάνω και με άλλους τέτοιους οργανισμούς. Είναι σημαντική η συνεργασία με την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Εγώ πιστεύω ότι δεν εκτιμούμε αρκετά το έργο των οργανισμών πάντοτε. Είναι σημαντική για το έργο και της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Εγώ είμαι και σκιώδης των ε, σοσιαλιστών για τον οργανισμό δεδομένων και πάντοτε θέλω να μιλάω για τη σημασία των οργανισμών γιατί πολλοί ε, πιστεύουν ότι οι οργανισμοί συνεπάγονται μόνο κόστη χωρίς να έχουν καλές επιδόσεις, ενώ ισχύει το αντίθετο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως το έκανε και στο παρελθόν, θα πρέπει να ενισχύσει το έργο των οργανισμών. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να προοικοδοτηθούν και αναλόγως από τον προϋπολογισμό και από τους ίδιους πόρους. Και αυτό είναι ένας τομέας πρέπει να το τονίζουμε πάντοτε. Δεν γίνεται οι οργανισμοί να παίρνουν και άλλα καθήκοντα χωρίς να έχουν πόρους και ανθρώπινους πόρους. Ε, υπάρχουν ε, προτάσεις για πιθανές συγχωνεύσεις, παύσεις, λειτουργίας ή και η μεταβίβαση καθηκόντων στην Επιτροπή. Αυτό μου δημιουργεί μια κάποια δυσαρέσκεια, ιδιαίτερα ε, το ερώτημα αν όλοι οι οργανισμοί χρειάζονται θα πρέπει να ε, παρακολουθούνται από το ελεγκτικό συνέδριο. Είναι πολύ σημαντικό το έργο τους, το έργο τους και χαίρομαι για την, τον ετήσιο, την ετήσια έκθεση για την διαχείριση και τον έλεγχο των ε, οργανισμών. Το δίκτυο των οργανισμών είναι πολύ σημαντικό και ο συντονισμός των οργανισμών ε, έχει έτσι βελτιωθεί και συνεργασία τους. Στο σημείο 3 ίσως θα έπρεπε να ε, διευκρινίσουμε ε, λίγο το θέμα, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Τσέλερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι Σκιώδη είναι ο συνάδελφος Σάουερμαν, ο οποίος σήμερα δυστυχώ δεν μπόρεσε να έρθει και γι' αυτό με παρακάλεσε να διαβάσω μια σύντομη ε, τοποθέτηση. Ή θέλει να ζητήσει συγγνώμη που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και ευχαριστεί τον κύριο Ντεγιόν για το σχέδιο γνωμοδότηση. Ο κύριο Σάουερμαν. συμφωνεί και στηρίζει την θέση του εισηγητή στη γνωμοδότηση, του συντάκτη τη γνωμοδότησης και θέλει να θέσει τρία θέματα ακόμη. Ε, Συντελεστέ θα πρέπει να ε, διορθωθούν για να αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος. Οι προπολογισμοί των οργανισμών θα πρέπει να ετοιμάζονται σύμφωνα με την αρχή του προπολογισμού βάση επιδόσεων και τρίτον μια θεματική προσέγγιση ε, στους οργανισμούς χρειάζεται για καλύτερη ιεράρχηση των καθηκόντων των οργανισμών, αυξημένη ε, συνεργασία, μειωμένη επικάλυψη, ιδιαίτερα σε οργανισμούς που εργάζονται και δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του ιδίου τομέα πολιτικής. Ευχαριστώ. Μία πρόταση που είναι σημαντική για μένα. Ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε καμία γνώμη στη μεταγκατάσταση της ΕΜΑΕΗ, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμού, είναι απαράδεκτο και δεν θα πρέπει να επαναληφθεί στο μέλλον. Ναι, πολύ ασχοληθήκαμε με τους οργανισμούς και εγώ πέντε χρόνια εργάστηκα στην ομάδα εργασίας και τα έγγραφα ήταν τόσο μεγάλα που έπρεπε να κουβαλάει κανείς μπαούλα για να τα μεταφέρει. Κάναμε πολλά. Ε, προσπαθήσαμε πολύ, αλλά δεν βγήκε κανένα καλό αποτέλεσμα. Γι' αυτό καλό θα ήταν να, να ε, τα καταφέρουμε αυτή τη φορά καλύτερα. Έχετε το λόγο κύριε Γενική Γραμματέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν Ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω πως συμφωνώ με κάποιε από τι παρατηρήσει που έγιναν και από εσά και από τον εισηγητή και από τα μέλη της Επιτροπής αυτής, αλλά δεν θα έλεγα πώ δεν έχει γίνει τίποτα ή δεν έχουμε πετύχει τίποτα μέχρι τώρα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, αποδοτικότητα εμείς εκμεταλλευόμαστε αυτή τη στιγμή με την αποδοτικότητα πολύ καιρό πριν μπουν οι συστάσεις ε, των διοργανικών επιτροπών για τις ε, υπηρεσίες και το έχουμε κάνει αυτό με αξιοσημείωτο τρόπο, δηλαδή αποδοτικότητα στη ε, χρήση των υπηρεσιών πληροφορικής, στις κρατικές προμήθειες, στις λογιστικές υπηρεσίες που προμηθευόμαστε και άλλες. Να δώσουμε λοιπόν το μήνυμα όπως το λαμβάνουμε δεόντως υπόψη και θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε κατά πόσο υπάρχει και περιθώριο για περισσότερη αύξηση της αποδοτικότητας. Να σας πω το εξή όμω. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για να συγχωνευθούν δύο υπηρεσίες, δεν τα κατάφερε, αποτύχαμε παταγωδός και θα πρέπει να καταθέσουμε νέα πρόταση. Ε, δεν μπορούμε εμείς να συγχωνεύουμε μόνο και μόνο για να συγχωνεύουμε. Οι υπηρεσίες όσους έχουν σήμερα έχουν διαφορετικές εντολές. Μπορούμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε στο Παρίσι, ας πούμε, ε, όπου θα πάει η, η έμπα μετά το ε, Λονδίνο και κάποια άλλα θέματα, αλλά δεν μπορεί απλώς κανείς να συγχωνεύει απλώς για να έχει μικρότερο ρυθμό υπηρεσιών όταν έχουν τελείως διαφορετικές εντολές. Κάποιοι από εσά μιλήσατε για την ε, μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων από το Λονδίνο. Ξέρετε ποια είναι τα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Μητροπή δεν είναι μεγάλος παίκτη στο θέμα αυτό είναι θέμα μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Γιατί η πρακτική εδώ και δεκαετίες είναι να αποφασίζουν τα κράτη-μέλη το θέμα του, της έδρας των υπηρεσιών. Και τώρα βέβαια υπάρχουν κάποιες ε, φωνές που ζητούν να αλλάξει αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μία θεσμοθετημένη διαδικασία και νομίζω ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να το δουν και καλό ήταν να δούμε τι έγινε με την ΕΜΠΑ, την Τραπεζική ε, Υπηρεσία και τον Οργανισμό Φαρμάκων ε, για το πώς θα εγκατασταθούν αυτές σε άλλες πρωτεύουσες και μέχρι τον Απρίλιο θα σας έχουμε δώσει και μία έκθεση με τα αποτελέσματα τα δικά μας αλλά δεν μπορούμε εμείς να προδικάσουμε τι θα γίνει με το μελλοντικό καθεστώς ή με τις μελλοντικέ πρακτικές. Αυτό θα πρέπει να το επαναδιαπραγματευτούν τα τρία θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλά, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Και ο εισηγητής για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, ε, δεν είναι όλοι ίδιοι. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς ε, επιτελούν εξαιρετικό έργο. Αυτό θα πρέπει να το πούμε πιο καθαρά ίσως στην εκθεσή μου. Δεν αναφέρω ότι είμαστε ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους. Θα μπορούσαμε να το λέμε πιο καθαρά και να πούμε ότι είναι και σημαντικό το έργο τους επίσης. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Σαββάνα, με όλα τα σημεία. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε κάποιες προσθήκες, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι στη δεύτερη διοργανική ομάδα εργασία, στην οποία εγώ συμμετείχα ως εκπρόσωπος της Επιτροπής μας, εκεί η Επιτροπή ουσιαστικά δεν λέει ποτέ αυτά που είπε εδώ η Επιτροπή θα κάνει πολύ καλή δουλειά και όταν μιλάμε για οργανισμούς έχουμε τον οργανισμό για τους Ιδεροδρόμους που βρίσκεται σε δύο τοποθεσίες μέσα στο ίδιο κράτος μέλος. Τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά εδώ και καιρό και ακόμα δεν έχουμε λάβει διευκρινήσεις για το ποιος είναι ο λόγος που δεν υπάρχει απλά μία τοποθεσία. Επίσης, ε, μερικές φορές έχουμε μία εντολή και δύο οργανισμούς που θα μπορούσαν να συγχωνευθούν. Σίγουρα από πολιτική άποψη είναι δύσκολο. Αλλά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν την έχουμε για να μας λέει ότι κάτι είναι δύσκολο. Αν είναι να υπερασπίζεται την αποτελεσματικότητα. Τι σημασία έχει πόσο δύσκολο είναι πολιτικά. Ο κ. Τίμερμανς έχει ξεκινήσει τις εργασίες, αλλά όπως φαίνεται προς αυτή την κατεύθυνση δεν υπάρχει ιδιαίτερη πρόθεση να επιτευχθούν αποτελέσματα. Είναι απαράδεκτο αυτό. Κανείς δεν φαίνεται να θέλει να γίνει ούτως ή άλλως. Κοιτάξτε, αυτή την πρόταση της Κομισιόν την στηρίξαμε για την συγχώνευση των οργανισμών, μην νομίζετε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Και είχαμε και ιδέες σχετικά. Πάμε στο επόμενο το και τελευταίο. Μια μελέτη. Ο κύριος Μπλόμαϊερ είναι πάλι εδώ. Συγγνώμη που περιμένατε, αλλά σήμερα είχαμε μια καθυστέρηση. Έχετε το λόγο για να κάνετε την παρουσίαση της μελέτης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ζήτησε ο κύριος De να έρθουμε και να το παρουσιάσουμε. Είναι μια ενημέρωση. Δεν είναι πλήρης μελέτη, είναι ενημέρωση. Κάτι διαφορετικό από αυτό που έχετε συνηθίσει. Αλλά ακολουθεί μετά από μια μελέτη που σας καταθέσαμε το 2015 και η οποία εξέτασε τι γίνεται με το μητρό των εμπειρογνωμόνων. Ξέρετε πως έκτοτε έχουν συμβεί πολλά. Οπότε μας ζήτησαν να το ξαναδούμε. Το κάναμε το καλοκαίρι φέτος. Και είδαμε και την ποσοτική ενημέρωση και αξιολόγηση χρησιμοποιώντας τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το μητρό της. Τα επεξεργαστήκαμε, και στείλαμε και ένα ερωτηματολόγιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας ευχαριστώ κύριε Κλάους που μας δώσατε πολλές απαντήσεις και λεπτομέρειες. Um, present, um, yeah, some of the sort of um, key, key data. Κάποια λοιπόν από τα κομβικά συμπεράσματα για το σύστημα αυτό των εμπειρογνωμών τα είδαμε και εστιάσαμε σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία προκάλεσαν όντως ανησυχία. Στην προηγούμενη έκθεση του 2015, δηλαδή η διαφάνεια, η ισορροπία και προσθέσαμε εδώ ένα νέο θέμα το οποίο δεν είχαμε εξετάσει το 2015 που είναι το φύλλο, η ισορροπία δηλαδή μεταξύ των δύο φύλλων. Για να δούμε λοιπόν γιατί έγινε αυτή η μελέτη και η προηγούμενη, πρέπει να σας πω πως εγώ στο Exeter διδάσκω πολιτικές επιστήμες και πρόσφατα είδα, βρήκα ένα ε, συγγράμμα το οποίο εξέταζε το θέμα αυτό των ομάδων εμπειρογνωμόνων και του Μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το συνέκρινε με αντίστοιχα συστήματα στα κράτη-μέλη. Να σας διαβάσω, να σας το παραθέσω για τις επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ευνοϊκό καλοήθες ε, περιβάλλον ε, που εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα και γίνεται εκεί και μια σύγκριση με τα ευρωπαϊκά κράτη και λέει ότι μπορούν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, και άλλες ομάδες να παραμείνουν εκτός διαδικασίας. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ επικριτικό και σίγουρα στο σωστό πλαίσιο θα πρέπει να το δούμε γιατί είναι μια δήλωση η οποία βασίστηκε σε κάποιες ε, ε, ε, εξετάσεις που έγινε του συστήματος πριν την αναθεώρηση του 16 και όπως γνωρίζετε κι εσείς μετά το, τις δράσεις του διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το σύστημα αυτό των εμπειρογνωμών αναθεωρήθηκε το Μάιο του 2016 και λάβαμε νέου οριζόντιου κανόνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού βρισκόμαστε τώρα, Ιούλιο του 18. Εκεί κοιτάξαμε το σύστημα μέσω της βάσης δεδομένων. Λοιπόν, στο πρώτο διάγραμμα βλέπετε τους συνολικούς αριθμούς, τα θρίσματα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 15.515 μέλη 700, 755 ομάδες. Βλέπετε λοιπόν ε, τι γίνεται σε αριθμό μελών από τότε. Έχουμε ε, λιγότερο μεγάλη μείωση των ε, ειδικών, αλλά έχουμε από 24.788 από 788-755 το, το 15 μέχρι το 18. Και μετά το 2006 είχαμε 1.300 ομάδες εμπειρογνωμόνων, ε, δηλαδή η καθοδική πορεία συνεχίστηκε. Εδώ έχουμε μια σύγκριση μεταξύ 2015 και 2018 για στις πέντε κατηγορίες. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν διάφορα είδη εμπειρογνωμόνων αυτοί που λειτουργούν υπό την ατομική τους ιδιότητα διότι έχουν συγκεκριμένες γνώσεις, συγκεκριμένο κύριο σε ένα τομέα και άλλοι που εκπροσωπούν κάποια συμφέροντα και για τις δύο αυτές ομάδες ε, έχουμε κάποια νούμερα και για τις μεγάλες, μεγαλύτερες ομάδες για οργανισμούς, για κρατημέλη έχουμε σημαντική μείωση στα μέλη μεταξύ αυτών των δύο ετών και έχουμε μια νέα κατηγορία που δεν υπήρχε το 2015 την εισήγαμε τους νέους οριζόντους κανόνες. Λυπή. Από όσο θυμάμαι, μιλάμε για οργανισμούς τρίτων χωρών, οργανισμούς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μόλις αναφέραμε και άλλων ειδών διεθνείς οργανισμοί που στο παρελθόν αποτελούσαν κομμάτι των οργανισμών, αυτής της κατηγορίας των οργανισμών. Τώρα, από μια άλλη οπτική γωνία, αν δούμε τα μέλη το 2018, εδώ σε αυτό το διάγραμμα τι προσπαθούμε να σας δείξουμε με πορτοκαλί χρώμα βλέπετε σαφώς ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των μελών προέρχονται από τα μελή, εκπρόσωποι των κρατών μελών και μικρότερα μερίδια οι ατομικοί, οι επιμέρους εμπειρογνώμονες, ε, οι λοιποί και 23% περίπου οι οργανώσεις. Κάτι σημαντικό θα θυμάστε ε, και συζητήθηκε και στη μελέτη του 2015 είχαν εκφραστεί επικρίσεις στο παρελθόν από τους οργανισμούς ε, της κοινωνίας των πολιτών ότι δεν ήταν πάντα σαφές ε, ποιον εκπροσωπούν εκπρόσωποι ουσιαστικά των κρατών μέλων και ποιοι ήταν. Και αυτοί οι νέοι οριζόντιοι κανόνες του 2016 κατέστησαν σαφές ότι οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών πρέπει να είναι δημοσιοί οι εκπρόσωποι του δημοσίου, υπάλληλοι του δημοσίου. Αν πάμε εδώ τώρα στους οργανισμούς πιο συγκεκριμένα, διότι αυτή η κατηγορία έχει γεννήσει κάποιες ανησυχίες στο παρελθόν, εδώ στο διάγραμμα βλέπουμε σαφώς την προέλευση. Όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών συμφερόντων ή επιχειρησιακών και μη επιχειρησιακών συμφερόντων, αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Οπότε βλέπετε εδώ υπάρχουν πολλές κατηγορίες ενός επαγγελματιών, ε, επιχειρήσεων, συνδικάτων, τράπεζες, ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ε, δικηγορικές εταιρείες, συμβουλευτικές εταιρείες, πολλές υποκατηγορίες δηλαδή, που σχετίζονται με κάποια οικονομικά ή επιχειρηματικά συμφέροντα και άλλες με μη οικονομικά συμφέροντα, μη επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχουμε ΜΚΟ που αποτελούν το 2% για παράδειγμα. Για κάποιους τομείς εστίασης τώρα της μελέτης, ε, η εξισορρόπηση μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών συμφερόντων και εδώ οι οριζόντιοι κανόνες του 2016 είπαν πολύ ρητά ότι υπάρχει δέσμευση για ισορροπημένη σύνθεση. Ήδη στι εισαγωγικέ αιτιολογικέ σκέψει θεσπίζεται αυτή η αρχή. Ωστόσο, όπω γνωρίζετε επίση, δεν πάβει να αποτελεί στόχο που έχει οριστεί και που δεν έχει ακόμα στόχο ουσιαστικά για την επίθεση κάποιου είδους ισορροπία. Τώρα, προσπαθήσαμε να επαναλάβουμε το εγχείρημα του 2015 για να δούμε στις ομάδες εμπειρογνωμόνων όπου εκπροσωπούνται οικονομικά συμφέροντα πώς έχουν τα πράγματα. Υπάρχει καλή εξισορρόπηση. Και τα στοιχεία μας μας λένε ότι ενώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, εξακολουθούμε να παρατηρούμε ότι στο 75% ή στο 74% των ομάδων εμπειρογνωμόνων, όπου έχουμε μέλη οικονομικών συμφερόντων, αυτοί αποτελούν την πλειοψηφία. Στο 20% των ομάδων τα πράγματα είναι αντίστροφα. Εάν είναι πλειοψηφιακή τα μη οικονομικά συμφέροντα και στους 6% έχουμε ισορροπία. Τώρα, εδώ ουσιαστικά ίσω να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φανταστείτε, εδώ έχουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με κάποια μέλη οικονομικών συμφερόντων, μη οικονομικών συμφερόντων. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα εδώ, διότι το θα ακουστούν τα μη οικονομικά συμφέροντα. Εδώ κάναμε κάτι άλλο. Το είχαμε κάνει ήδη το 2015. Κοιτάξαμε το βαθμό ανισορροπίας. Ε, υπάρχουν διάφορε κατηγορίε εδώ. Έχουμε την κρίζα κατηγορία 7% που δεν υπάρχει έλλειψη ισορροπίας. Ε, είναι η ισορροπία μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών μελών. Με κίτρινο το 22% εδώ έχουμε πολύ χαμηλή διαφορά. 0,25 κάτω από το 0,50% των μελών. Έχουμε τη μεσαία κατηγορία σχεδόν 50% όπου περίπου το 1 τέταρτο των μελών των ομάδων εμπειρογνωμών εκπροσωπούν τα μη οικονομικά συμφέροντα και μετά έχουμε την πιο ανησυχητική κατηγορία που παρουσιάζει τεράστια έλλειψη ισορροπίας, ομάδες εμπρογνωμόνων όπου τα μέλη οικονομικών συμφερόντων είναι παρόντα μεν, χωρίς ε, να υπάρχουν μέλη που, δεν εκπροσωπούν, μη που εκπροσωπούν μη οικονομικά συμφέροντα. Και πάλι αυτό αποτελεί τεράστια βελτίωση σε σχέση με τα στοιχεία του 2015. Τότε δεν ήταν 23% το ποσοστό, αλλά 72%. Αυτές οι ομάδες εμπειρογνωμόνων με απουσία εκπροσώπησης των μη οικονομικών συμφερόντων. Πάμε στη δεύτερο τομέα εστίαση, στη διαφάνεια. Και εδώ έχουμε πολλές καινοτομίες στο πλαίσιο οι δημόσιες ε, ε, προσκλήσεις υπάρχουν ε, που αποτελούν τον κανόνα, δεν υπάρχουν χωρίς εξαιρέσεις. Ξέχασα να σας αναφέρω επίσης ότι υπάρχει μια σημαντική σύνδεση τώρα μεταξύ του Μητρώου Ομάδων Εμπειρογνωμόνων και του Μητρώου Διαφάνειας. Αυτό επηρεάζει του εμπειρογνώμονε που εκπροσωπούν συμφέροντα και του οργανισμού που πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρό Διαφάνεια για να είναι επιλέξιμε για συμμετοχή στι ομάδε εμπειρογνωμόνων. Και πάλι αυτό το χειριζόμαστε με μεγάλη αυστηρότητα όπως δείχνουν τα στοιχεία διότι η Κομισιόν έχει παράσχει ε, πληροφορίες για μεγάλο αριθμό 120 μέλη έχουν ε, αποκλειστεί γιατί δεν πληρούσαν αυτή την προϋπόθεση. Κάτι άλλο σημαντικό καινούριο ε, υπάρχει η σύγκρουση συμφερόντων για επιμέρους ε, μέλη. Πρέπει να υποβάλουν μια δήλωση συμφερόντων και να δηλώνουν τις σύγκρουσεις συμφερόντων και τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό εφαρμόζεται. Γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των αιτήσεων που απορρίφθηκαν ουσιαστικά λόγω διαπίστωσης σύγκρουση συμφερόντων. Έχουμε την αίσθηση παρόλα αυτά ότι παρότι οι πρόοδοι είναι σημαντικέ όσον αφορά την πρόσβαση στι προφορίε και στα όσα συμβαίνουν, στι ομάδε εμπειρογνωμόνων, στα έγγραφα που παράγουν, ε, υπάρχει διαθεσιμότητα στις ιστοσελίδες του συνήθως. Ε, Παρ' όλα αυτά, Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ομάδες εμπειρογνωμόνων αποφασίζουν να μην δημοσιοποιήσουν κάποια έγγραφα. Και επίσης έχουμε παρατηρήσει ότι ελάχιστε ομάδες εμπειρογνωμόνων, μόνο 12 έχουν ανοίξει τις ε, συναντήσεις τους ε, για το κοινό ή χρησιμοποιούν το web streaming για την κοινοποίηση των πληροφοριών. Uh, um, Ο τελευταίος τομέας εστίασης που εξετάσαμε είναι η ισορροπία μεταξύ των φύλων. Ε, κάτι καινούριο επίσης. Με τους νέους οριζόντους κανόνες του 2016 εισηχθεί στόχος ε, τουλάχιστον 40% για την εκπροσώπηση κάθε φύλου ε, στις ομάδες και βάσει των βάσεων δεδομένων μας ε, από τις 129 ομάδες, ε, στις 129 ομάδες ακόμα δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος. 107, σε 107 ομάδες αυτό αφορά γυναίκες, όπου δεν επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος του 40%. Και για 22 ομάδες ε, δεν επιτυγχάνεται ο στόχος για τους άρενες εκπροσώπους. Πολύ γρήγορα τώρα οι συστάσεις. Τι κάναμε στο πλαίσιο τη μελέτη. Επίσης, ξαναείδαμε όλες τις συστάσεις που είχαμε εκδώσει και υποστηρίξει ε, στην Επιτροπή το 2015. Κάποιες εξακολουθούν να ισχύουν, πιστεύουμε. Και πιστεύουμε ότι αυτή, αυτός ο ποσοτικός απολογισμός θα μπορούσε να μας βοηθήσει να δούμε τι θα κάνουμε με τα υπόλοιπα ζητήματα. να δούμε πιο συγκεκριμένα με αυτές τις 39 ομάδες εμπειρογνωμών που θεωρούμε ότι χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό ε, ανισορροπίας για να δούμε ουσιαστικά πώς ε, τα μέλη που εκπροσωπούν με οικονομικά συμφέροντα θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις ομάδες να συμμετέχουν ή να ε, καταφέρουν να ακουστεί η φωνή τους σε αυτές τις ομάδες. Επίσης θα μπορούσαν να γίνουν και περισσότερα για την άνοιγμα στο κοινό των συναντήσεων, να μειωθούν οι εξαιρέσεις στη δημοσιοποίηση των εγγράφων και φυσικά να ε, βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ της εκπροσώπησης των φύλων. Τέλος, ε, κάναμε μία αναθεώρηση των ομάδων για να δούμε αν έχει κυκλοφορήσει κάτι καινούργιο στη βιβλιογραφία όσον αφορά τις ομάδες εμπειρογνωμόνων από την τελευταία φορά που το είχαμε κοιτάξει. Μας έκανε έκπληξη ότι βρήκαμε ελάχιστα πράγματα. Όπως ξέρετε, αυτή η διαδικασία έγινε μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Περισσότερο ποιοτικά, ποσοτικά, οι αριθμοί δεν μας δείχνουν αρκετά τις εξελίξεις. Θέλαμε να γίνει μια έρευνα σε μεγαλύτερο βάθος ενδεχομένω εσωτερικά από την Κομισιόν κάποιε αξιολογήσει τη απόδοση του συστήματο των ομάδων εμπειρογνωμών. Ευχαριστώ. thank you very much. We need to continue without interpretation in Ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε με τα αγγλικά χωρίς διερμηνία. Παρακαλώ, κύριε Σαγητά. and uh, also a big thank you to uh, um, the researcher and uh, the researchers, Mr. Blomeyer, also for his presentation of the research.